Κύριε Πρόεδρε, καλωσορίσατε στην τελευταία αυτή ανταλλαγή απόψεων στα πλαίσια του νομισματικού διαλόγου στη διάρκεια αυτής της θετίας του Κοινοβουλίου. Στα πέντε χρόνια που πέρασαν είχαμε μια πολύ καλή συνήθεια η οποία βελτιώνεται με τα χρόνια. Βέβαια πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν προκειμένου οι ανταλλαγές αυτές να, γι... να βιώνονται και να γίνονται κατανοητές μες στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου στο σωστό ύψος σε αυτό που επιβάλλετε. Αλλά όταν εσείς ως πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας έρχεστε να κάνετε μια, ένα απολογισμό της δραστηριότητας της Κεντρικής Τράπεζας και να μας παρουσιάσετε την στρατηγική την οποία εφαρμόζεται προκειμένου να φέρετε σε πέρα στην αποστολή που σας ανέθεσαν οι συνθήκες. Για την τελευταία αυτή λοιπόν ανταλλαγή απόψεων επιλέξαμε δύο θέματα. Οι συνέπειες για την ευρωζώνη της σημερινής κρίσης και ο ρόλος της κεντρική Τράπεζας στην εποπτεία των χρηματαγορών. Βέβαια, για το δεύτερο θέμα, η δημοσίευση της έκθεσης Λαροζιέρα και εμείς θα έχουμε μια ακρόαση για το θέμα αυτό στις 23 Απριλίου έχει ιδιαίτερη σημασία ε, και τα μέλη της ε, τράπεζας εξέφρασαν θέσεις σχετικά με το ρόλο της κεντρικής τράπεζας όσον αφορά την εποπτεία. Θα μας ενδιαφέρει όμως να ακούσουμε την άποψή σας και την αξιολόγησή σας σχετικά με το τι θέση πρέπει να πάρουμε μεταξύ του επίγοντος χαρακτήρα, οι άμεσα μέτρα δράσης και από την άλλη μεριά την ανάγκη μια ευρωπαϊκού επίπεδου εποπτείας. Αμέσω σα δίνω το λόγο χωρί καθυστέρηση και μετά όσοι ήθεστε, θα περάσουμε στι ερωτήσει και τι απαντήσει. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία, κυρία Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι ευρωβουλευτέ μέλη τη Επιτροπή Νομισματικών Θεμάτων, χαίρομαι που για τρίτη φορά ε, παρουσιάζομαι στο Ευρωκοινοβούλιο να μιλήσω δεύτερη φορά στην Επιτροπή σα. Επίση, δεν ξεχνάω και την κοινή συνάντηση που είχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα Εθνικά Κοινοβούλια το Φεβρουάριο. Τέσσερις φορές λοιπόν συνολικά με διαφορετικές μορφές ήρθα, έχω έρθει στο κοινοβούλιο. Η σημερινή συνάντηση όπως είπατε είναι η τελευταία που προβλέπετε για την πενταετία αυτή. Έχει ιδιαίτερη σημασία όπως είπατε και επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω ήδη για τις πάρα πολύ πλούσια ανταλλαγή απόψεων που είχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Είναι η 21η φορά ακρόαση για μένα στην Επιτροπή Νομισματικών Θεμάτων, πράγμα το οποίο μαρτυρεί την στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και των εκλεγμένων εκπροσώπων της Ευρώπης, όπως πολύ σωστά το είπατε. Σήμερα θα ήθελα να αναφερθώ σε τέσσερα θέματα. Η τρέχουσα οικονομική κατάσταση, η δομή χρηματοδότησης ιδιωτικών ακινήτων στην Ευρωζώνη, οι επιπτώσεις της κρίσης σε μια μελλοντική εισαγωγή στο ευρώ των κρατών μελών της ε, κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και τέταρτο, οι προτάσεις για μεταρρύθμιση του συστήματος εποπτείας στην Ευρώπη. Ελπίζω ότι έτσι ε, θα αναφερθώ σε μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα. Πριν φυσικά όσοι ήθεστε θα είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Συνεχίζει στα αγγλικά. Θα αρχίσουμε την οικονομική κατάσταση και τις πρόσφατες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής. Σημειώστε, και το ξέρετε βέβαια, ότι τρεις μέρες πριν την επόμενη συνάντηση νομισματικής πολιτικής, την Πέμπτη, βρίσκομαι στην φάση πέρντα, όπως τη λέμε, και θα παραμείνω σε αυτή την στάση, φάση, γιατί ε, δεν, υποτίθεται δεν μπορώ να πω τίποτε το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει τι αποφάσει αυτή τη εβδομάδα. Από τότε που μίλησε στο Ευρωκοινοβούλιο την τελευταία φορά στι 21 Ιανουαρίου, η οικονομική κατάσταση και η προοπτική τη ε, εξασθένησαν περαιτέρω. Οι πληθωριστικέ πιέσει μειώθηκαν, όπω επιβεβαιώνεται αυτό από τι τάσει του μισματικού και πιστοτικού χαρακτήρα του Φεβρουάριου. Το Φεβρουάριο ο πληθωρισμό ήταν χαμηλό, γύρω στο 1,2% και όπω ξέρετε η μείωση στον πληθωρισμό από πέρυσι το καλοκαίρι κυρίω αντικατοπτρίζει την μεγάλη μείωση των τιμών πρώτων υλών. Με προοπτική ε, αναμένουμε ο πληθωρισμός να είναι αρκετά κάτω από το 2% για φέτος και το 2010. Ο κίνδυνος αυτής της προοπτικής είναι σχετικά ισορροπημένος και χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας. Μετά την εξασθένιση της παγκόσμιας οικονομίας, μετά την χρηματοπιστωτική θύελα, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ευρωζώνη μειώθηκε πάρα πολύ, κατά 1,5% ανά τρίμηνο, στο τέταρτο τρίμηνο του 2008. Οι τελευταίες πληροφορίες μας λένε ότι η οικονομική δραστηριότητα επιδεινώθηκε περαιτέρω το πρώτο τρίμηνο του 2009. Η ζήτηση θα παραμείνει ασθενής για όλο το 2009 και σε συνολικό επίπεδο και στην Ευρωζώνη πριν βαθμία ανακάμψη το 2010. Όπως συμβαίνει και με τον πληθωρισμό, αυτή η προοπτική επίσης χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Κίνδυνος για αυτή την προοπτική φαίνεται να είναι κάπως πιο ισορροπημένος. Από τη μια μεριά, η θετική επίπτωση των πρόσφατων πακέτων διάσωση εκ μέρου των κυβερνήσεων για τις τράπεζες και ο μακροοικονομική τόνωση η οποία αυτή τη στιγμή υλοποιείται ίσως είναι πιο ισχυρή από ό,τι προβλεπόταν. Από την άλλη μεριά η επίπτωση της χρηματοπιστωτικής θύελας που συνεχίζεται επί της πραγματικής οικονομίας είναι πιο ισχυρή από ό,τι το Επιπλέον ε, δημιουργούνται προστατευτικέ τάσει που δημιουργούν ανησυχία. Με όλα αυτά τα δεδομένα η το Διοικητικό Συμβούλιο μείωσε κατά επιπλέον 500 βασικά σημεία στις αρχές Μαρτίου το επιτόκιό μας. Οπότε η συνολική μείωση ήταν κατά 275 σημεία βάσης από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα. Συνολικά η σταθερότητα των τιμών πιστεύουμε ότι θα διατηρηθεί μέσω πρόθεσμα. Θα συνεχίσουμε να τηρούμε την εντολή που μας δόθηκε να συνδέουμε τις προσδοκίες πληθωρισμού με μακροπρόθεσμη διάσταση. Αυτή η σύνδεση για βιώσιμη, ε, συμβάλλει σε βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση και επίσης σε χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Επίσης σας θυμίζω ότι η Κεντρική Τράπεζα προσάρμοσε το πλαίσιο διαχείρισης της ρευστότητα προκειμένου να καλυφθούν οι δυσλειτουργίες στην ε, Ευρωζώνη όσον αφορά τις χρηματαγορές. Το πιο σημαντικά μέτρα ήταν τον Οκτώβριο του 2008 όπου, ισχύει, ε, όπου οι διαδικασίες δημοπρασιών με σταθερό επιτόκιο ε, και για μεσοπρόθεσμες και για μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις εισήχθη, όπως επίσης η επέκταση μέχρι το τέλος του 2009 ενός καταλόγου επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού για χρήση ως εγγύηση, collateral, σε ε, πράξεις πίστοσης στην Ευρωζώνη αποφασίσαμε τη διαδικασία αυτή να διατηρηθεί όσο χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει και πέραν του τέλους του 2009. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των μέτρων, ε, τα περισσότερα από τα οποία δεν είναι στάνταρ, οι τράπεζες εξακολούθησαν να έχουν ευρεία πρόσβαση στην ευρωρευστότητα. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο θέμα. Η χρηματοδότηση κατοικιών που υπάρχει και στην έκθεση διαθροτικών θυμάτων της έκθεσης. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια θα σα παρουσιάσω τις γενικές γραμμές της έκθεσης, η οποία θα δημοσιευθεί σήμερα προς το τέλος τη ημέρα. Η έκθεση αναλύει τάσεις και διαφορές στα χαρακτηριστικά των στεγαστικών δανείων, στην χρηματοδότηση τραπεζικών δανείων και στη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των επιτοκίων ε, των δανείων και στο κόστος χρηματοδότησης των τραπεζών. Όπω επίση λαμβάνεται υπόψη το τι συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Γενικά, οι τράπεζε στην Ευρωζώνη είναι πολύ πιο αυστηρέ όσον αφορά του όρου εκτό επιτοκίου επί των δανείων. Αυτό εν μέρη εξηγεί το ότι ε, ο τομέας των subprime είναι πολύ πιο μικρός εδώ. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, σχετικά σταθερές καταθέσεις τραπεζών εξακολουθούν η κύρια πηγή για τη χρηματοδότηση τραπεζικών δανείων στην Ευρωζώνη με λιγότερη έμφαση στην λειτουργία Originate to Distribute. Αυτέ οι παρατηρήσει υποστηρίζουν το συμπέρασμα ότι η, χρηματοδότηση, η στεγαστική χρηματοδότηση στην Ευρωζώνη ε, ε, είναι πιο ευέλικτη και αντέχει περισσότερο σαν αφορά τα σοκ. Η χρηματοδότηση στεγαστικών δανείων σαν επίπτωση στην νομισματική πολιτική επιδέχεται τα εξή δύο σχόλια. Πρώτον, ε, έχουμε πιο μεγάλο βαθμό ανταγωνισμού μεταξύ αυτών που παρέχουν αυτά τα δάνεια. Αυτό οδηγεί σε μια ενίσχυση αυτής της μεταβίβασης. Από την άλλη μεριά η εισαγωγή μεγαλύτερης ευελιξίας στα στεγαστικά δάνεια μέσω της προσωρινής άρσης των πληρωμών ή δανείων που έχουν λήξει θα οδηγήσει σε αλλαγές των επιτοκίων. Αυτό έχει μικρότερη άμεση επίπτωση στην οικονομία. Τέλος είναι σαφές ότι θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερο ποσοστό ε, κατακράτησης, retention, εκ μέρους των τραπεζών και όσον αφορά την ποσότητα και όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των δανείων που δίνονται στα νοικοκυριά όσον αφορά τις πηγές χρηματοδότησης. Ε, θα μπω τώρα στο τρίτο θέμα, τις συνέπειες της υφιστάμενης κρίσης σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση της ζώνης ευρώ. Η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινώθηκε ιδιαίτερα μετά το Σεπτέμβριο του 2008 συνέπεια της έντασης της χρηματοπιστωτικής κρίσεως. Κάποιες χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης επλήγησαν και αυτές σκληρά, υπογραμμίζοντας και ίδιο ακόμα περισσότερο παλαιότερες τροτότητες. Οι αδυναμίες αυτές σχετίζονται και με τις ε, έλλειψη ισορροπίας των χώριων και των εξωτερικών εμπόριο, την λανθασμένη φορολογική πολιτική και, την, ε, και το χρέος τους. Ωστόσο πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ των διαφορών χωρών στην περιοχή. Κάποιες χώρες έδειξαν σοβαρό βαθμό αντοχή σε, αυτή, σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Και δεν είναι περίεργο ότι οι χώρε που πλήγησαν περισσότερο από την κρίση είναι δυστυχώ εκείνε οι χώρε που είχαν δημιουργήσει μεγάλε ανισορροπίε και τροτότητε στο παρελθόν. Συνολικά, η, οικονομική κρίση έδειξε, η χρηματοοικονομική κρίση έδειξε τη σπουδαιότητα του να αποφεύγουμε μακροοικονομικές ανισορροπίες και να ακολουθούμε έναν δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης που υποστηρίζεται από ε, σοβαρό βαθμό διαθροτικών μεταρρυθμίσεων. Τούτο είναι ιδιαίτερα αληθές για οικονομίες που προσπαθούν να προλάβουν τις άλλες και που πρέπει να συνδυάσουν και την επιθυμία τους για γρήγορη σύγκληση και την ανάγκη να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα της διαδικασίας σύγκλησης. Η υιοθέτηση του ευρώ δεν μπορεί να είναι υποκατάστατο για την ανάγκη ε, προσαρμογής της εγχώριας πολιτικής, γιατί αυτό είναι κόντρα στην οικονομική λογική που στηρίζει και διέπει την διαδικασία σύγκλησης στην Ευρώπη και είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι η πρώιμη και πρόοριο θέτηση του ευρώ μπορεί να καταστήσει δυσκολότερο να μπορέσει μια χώρα να αντιμετωπίσει τις υπερχόμενες προκλήσεις. Χωρίς, την ε, χωρίς βιώσιμη σύγκληση η νομισματική πολιτική Τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να μην είναι ενδεδειγμένη για την συγκεκριμένη χώρα και σε μια τέτοια περίπτωση η χώρα αυτή θα μπορεί να αντιμετωπίσει μια, ε, μια ε, πτυτικότητα της, ε, του πληθωρισμού και να οδηγήσει σε έλλειψη οικονομικών σταθερών ε, συνθήκων στην πατρίδα. Η υιοθέτηση του ευρώ μπορεί να γίνει μόνο όταν υπάρχουν ε, δεν υπάρχουν πλέον μίζωνες ενισορροπίες στη χώρα και όταν ε, υπάρχει υπάρχει βιώσιμη σύγκληση όπως προβλέπει και η συνθήκη. Το τελευταίο θέμα τώρα που αναφέρατε πριν από λίγο κυρία Πρόεδρε, την αναθεώρηση του πλαισίου για την χρηματοοικονομική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φθινόπωρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών να παίξουν δραστήριο ρόλο στην ε, προληπτική εποπτεία σε μακροοικονομικό επίπεδο και την χρηματοοικονομική σταθερότητα. Ο ρόλο αυτό προβλέπεται και στην έκθεση τη ομάδα υψηλού επίπεδου υπό την παιδεία του κ. Ντελαροζιέρ. Καλωσορίζω τι προτάσει για την εποπτεία, την προληπτική εποπτεία σε μακροοικονομικό επίπεδο, ιδιαίτερα την δημιουργία ενό Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου υπό την, εποπτεία, υπό την αιγίδα του, της ΕΚΤ. Να τονίσω στους κάποιε παρατηρήσεις. Πρώτον, η, η, οι αποφάσεις και οι προτάσεις του Συμβουλίου αυτού θα, θα συμβάλλουν ε, στην, στην χρηματοοικονομική σταθερότητα της Ένωση, σύμφωνα με το σύστημα, με την έκθεση τη Ρωσία, θα εντοπίσει και θα εκτιμήσει κινδύνου και ιδιωτερότητες του οικονομικού σύστημα της κοινότητα, θα, θα προβλέπει, θα προειδοποιεί για κινδύνους και θα υιοθετήσει συστάσεις ε, πολιτική. Επίσης, η σύνθεση του συμβουλίου αυτού αντικατοπτρίζει την αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζουν οι κεντρικές τράπεζες στην προληπτική εποπτεία σε μακροοικονομικό επίπεδο. Τρίτον, το γεγονό ότι το ε, Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θα τεθεί ή υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών τραπεζών θα του επιτρέψει να εκμεταλλευτεί και την αναλυτική ικανότητα και την τεχνική υποδομή των κεντρικών τραπεζών στην ανάλυση τη νομισματική και χρηματοοικονομική σταθερότητας. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο θα χρειάζεται να επαφίεται σε ένα ευρύ φάσμα στοιχείων προληπτικής εποπτείας σε μάκρο και μικρο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι και η, Ευρωπαϊκή, και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των εποπτικών αρχών. Τέταρτον, για, το πλαίσιο, για να μπορέσει το πλαίσιο αυτό να λειτουργήσει όπως επιθυμούμε, είναι κρίσιμο οι προειδοποιήσεις κινδύνου να μετατρέπονται σε δράση, πολιτική δράση όσο, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται. Στο πλαίσιο αυτό το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου θα πρέπει να αναφέρει της να αναφέρει τους, τις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις που υιοθετεί στο Συμβούλιο Κοφίν. Επίσης θα πρέπει να παράσχουμε μια θεσμική βάση για την θέσπιση αυτού του Συμβουλίου και τι συναφής νέες αρμοδιότητες σε μακροοικονομικό επίπεδο προληπτικής ε, εποπτείας της, ε, της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κεντρικών Τραπεδών για να εξασφαλίσουμε και την ε, λογοδοσία και την νομική δυνατότητα. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στο πλαίσιο αυτό την ενεργοποίηση του, άρθρου 5 παράγραφος 6 της συνθήκης. Με, δεν θα μπορούσα να κλείσω τις σημερινές παρατηρήσεις μου κυρία Πρόεδρε χωρίς να σας ευχαριστήσω και εσάς κυρία Πρόεδρε και όλα τα μέλη της Επιτροπής για την τακτική ανταλλαγή απόψεων στην τελευταία πενταετία. Οι 21 ακροάσεις που προανέφερα απαιτέλεσαν σημαντικές ευκαιρίες για να λάβω προτάσεις και πληροφορίες από το μέλη του Κοινοβουλίου και Ψωνόματος, του Συμβουλίου των Διοικητών και του προσωπικού της Τράπεζας θέλω να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη προσοχή και την ε, συνεργασία σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τις εισαγωγικές παρατηρήσεις σας και τις εκτιμήσεις που, την εκτίμηση που δείξατε για το νομισματικό διάλογο. Έλεγα και εγώ στην εισαγωγή ότι οι διάδοχοί μας θα βελτιώσουν σίγουρα περαιτέρω το, την ποιότητα του διαλόγου αυτού, τόσο ώστε η κοινή γνώμη να έχει μεγαλύτερη επίγνωση ότι οι ανταλλαγές αυτές έχουν αποτελέσματα και ότι το θέμα της δημοκρατικής λογοδοσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υλοποιείται στην πράξη. Δίνω το λόγο κατευθείαν στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο Ζαν Πολ Γκοζές, μετά ο αντιπρόεδρος Γκασία Μαργκάγιο. 1,5 λεπτό. Κύριε Γκοζές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της ομάδας μας, σας ευχαριστώ για την επιμέλεια με την οποία ε, κινήθηκατε έναντι του Κοινοβουλίου και του νομισματικού διαλόγου και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η κυρία Πρόεδρος. Θα ήθελα να σα θέσω μια ερώτηση σχετικά με το ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την εποπτεία. Αναφερθήκατε σε αυτό. Θα μπορούσατε να μας πείτε πού βρίσκεται η προπαρασκευαστική φάση ε, δεδομένη της έκθεσης Τελαροζιέρ και θα σας κάνω και μια κάπως ε, ερώτηση αφθάδη. Μερικοί σχολιαστές λένε ότι για να έχουμε ανάκαμψη και να βγούμε πιο γρήγορα από την κρίση, πρέπει να δεχτούμε πληθωρισμό. Το ακούμε αυτό συχνά στο ραδιόφωνο, στι τηλεοράσει. Είναι ελκυστικό να λέμε αυτά τα πράγματα για τον πληθωρισμό. Γιατί παλιότερα ο κόσμο νόμιζε ότι κερδίζει έτσι και ότι ανεβαίνει η αγοραστική του δύναμη. Αυτή λοιπόν η ερώτησή μου η δεύτερη είναι κάπω πιο αυθάδη σε σχέση με την πρώτη. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα απαντήσω με τη σειρά. Για την πρώτη ερώτηση, όπως σας είπα και πριν, θεωρούμε ότι η λεωφόρος που ανοίγει η έκθεση Λαροζιέρ για την μακροπρονοητική εποπτεία αφορά και αυτή την Ήπειρο και την Αμερική είναι μια λειτουργία που δεν ήταν θεσμοθετημένη, παρότι ήταν σαφής, σαφές ότι είχε σχέση με την ευθύνη όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που καταρχήν έχει μια κεντρική τράπεζα είτε με βάση την εντολή που έχει πάρει είτε λόγω της φυσιολογικής της λειτουργίας να εξασφαλίζει την νομισματική σταθερότητα. Έχει ειδικέ ευθύνες και ειδικό όραμα λόγω αυτού. Φυσικά, το πάνω θα κρυθεί από την εφαρμογή. Είμαστε σε στενή επαφή με την Κομισιόν. Η Κομισιόν, η Επιτροπή, καλείται να κάνει προτάσεις. Υποθέτω ότι και εσείς είστε σε επαφή με την Κομισιόν. Αυτή θα γράψει τις προτάσεις. Έτσι ώστε με τις επαφές αυτές να διασφαλιστεί αυτή η λειτουργία να εφαρμοστεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Βέβαια μερικά ερωτήματα. Δεν θα ήθελα να προδικάσω την ανάλυση της Κομισιόν και της συνεργασίας που θα έχει με εμά. Πάντως, θεωρούμε σημαντικό ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι συστάσεις θα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση και στο σωστό λήπτη. Και θεωρούμε αποκηρούμε τον πρόεδρο του ΕΚΟΦΗΝ ότι αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία. Εξάλλου η Κομισιόν θα είναι παρούσα στο νέο αυτό συμβούλιο που δημιουργείται και θεωρούμε σημαντικό, όπως σας εξήγησα, να υπάρχουν όλα τα κατάλληλα input, υλικό που θα έρχεται, όσον αφορά την μακροπρονοητική εποπτεία όχι μικροπρονοητική. Η έκθεση Λαροζιέρ είναι σαφής. Εμείς εκφράσαμε την ε, θετική μας άποψη στο θέμα αυτό. Είμαστε θετικά διακείμενοι. Έρχομαι τώρα στην δεύτερη ερώτησή σας. Και εγώ έχω παραξενευτεί όπως και εσείς. Δεν είναι σαφές πουθενά από ό,τι ξέρω ότι η κεντρική τράπεζα δεν ενδιαφέρεται πια, δεν θα ενδιαφέρεται πια για τον πληθωρισμό στο μέλλον, τι συνέπεια θα είχε αυτό. Οι ίδιοι οι συμπολίτε μας θα διαπίστωναν ότι η κεντρική τράπεζα δεν ενδιαφέρεται την αγοραστική δύναμη του κοινού. Αυτό ήταν το πιο κακό Συνιάλο που θα μπορούσαμε να εκπέμψουμε προς τους συμπολίτες και τους καταναλωτές σε μια περίοδο όπου το πιο σημαντικό είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή. Οι χρήματα αγορές θα διαπίστωναν ότι με ορίζοντα το μεθεπόμενο μήνα θα είχαμε πληθωρισμό κάποια στιγμή και όλα τα, επιτόκια μέσω μακροπρόθεσμα αντί να είναι χαμηλά όπως είναι ευκταίο στις σημερινές συνθήκες, θα ανέβαιναν, γιατί θα ενσωμάτωναν αυτές τις πληθωριστικές προσδοκίες. Θεωρώ λοιπόν ότι και όσον αφορά την εμπιστοσύνη και όσον αφορά τη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας, αυτό που συζητιέται, και ξέρω όπως και εσείς ότι συζητιέται, είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να γίνει και το λέω με απόλυτη σαφήνεια. Στους, 329 εκατομμύρια συμπολίτε μας μέσω ημών ότι εμείς διασφαλίζουμε την σταθερότητα των τιμών μέσω μακροπρόθεσμα όπως το ορίζουν οι συνθήκες με τους συγκεκριμένους ορισμούς που έχουμε δώσει λιγότερο από 2% αλλά γύρω στο 2% μπορούν να υπολογίζουν σε μας. Αυτό θα το διασφαλίσουμε και επαναλαμβάνω σήμερα για την εμπιστοσύνη πρέπει σήμερα να πάρουμε τις κατάλληλες αποφάσεις σε όλους τους τομείς και στα νομισματικά. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό όλοι οι οικονομικοί φορείς και πιο συγκεκριμένα οι συμπογίτες μας να τους καθησυχάσουμε ως προς το ότι θα προστατεύσουμε μέσω μακροπρόθεσμα τη σταθερότητα των τιμών. Ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Τρισέ για τις 21 συναντήσεις που είχαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας και που θα συνεχιστούν και στην επόμενη. Έλεγε ο Σκαρουέλντ ότι δεν υπάρχουν θρασίες ερωτήσεις αλλά θρασίες απαντήσεις. Θα κάνω κι εγώ κάποια τέτοια ερώτηση. Πρώτον, στην τελευταία κοινή συνάντηση Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων καταλήξαμε στο συμπέρασμα ούτως ότι για να επιστρέψει η πίστη, να ξαναμπούν τα, οι και πρέπει να υπάρχει καθαρότητα στους ισολογισμούς, νέα στεγαστικά και καθαρισμός των ενεργητικών το σχέδιο του νέου Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ που δεν αλλάζει και πολύ από αυτό του Πόλσον ε, περιλαμβάνει ενίσχυση, αγορά των τοξικών ομολόγων από το δημόσιο. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε την, τις απαιτήσεις της για τις εγγυήσεις ε, ζητώντας ε, μεγαλύτερο ποσοστό ενεργητικού. Δεν υπάρχει κάποια αντίφαση στα δύο. Δεύτερη ερώτηση. Το ισπανικό τραπεζικό σύστημα φαίνεται ότι είναι φερέγγιο, έχει ρευστότητα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει υψηλό, υπάρχουν υψηλά επιτόκια, 50% ψηλότερα από άλλα κράτη. Πώς μπορεί να υπάρχουν υψηλά επιτόκια σε ένα καθαρό ένα σύστημα το οποίο έχει φερεγγιότητα και ρευστότητα. Ευχαριστώ. Όπως είπατε, τολμηρές ερωτήσεις θα έχετε, δεν ξέρω αν θα έχει, δεν πιστεύω να περιμένετε βέβαια, τολμηρή, αδιάκριτη απάντηση. Ξεκάθαρη απάντηση θα λάβετε. Για το πρώτο ερώτημα. Όπως ξέρετε, και στις δύο όχθες του Ατλαντικού υπάρχουν δυνατότητες και επιλογές αντιμετώπισης των τοξικών στοιχείων ή τόσο πάντων των δύσκολων στοιχείων των αγορών. Συνεργαστήκαμε με την Επιτροπή, προτείναμε κάποια στοιχεία που έλαβε υπόψη, κάποιες προτάσεις που έλαβε υπόψη η Επιτροπή, επιπρόσθετα των ε, επιλογών ανακεφαλαιοποίησης και εγγύσεων. Οι νέες αυτές επιλογές θα επιτρέψουν να διατηρήσουμε και να διαφυλάξουμε ε, ένα ισότιμο επίπεδο στην Ένωση. Να σας πω ότι με βάση τους δικούς μας υπολογισμούς μόνο στη ζώνη ευρώ τα κονδύλια των κινδύνων για τους φορολογούμενους είναι της τάξης του 23% του ΑΕΠ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 29% με βάση τα δικού τους δικούς τους υπολογισμούς. Εδώ συμπεριλαμβάνω τα πάντα και τις νέες επιλογές που αναφέρατε. Θα έλεγα ότι αυτό που είναι αναγκαίο τώρα δεν είναι να συσσωρεύουμε νέες αποφάσεις ή νέες δυνατότητες, αλλά να υλοποιούμε τις ήδη ληφθείς αποφάσεις, που είναι πολύ σημαντικές. Και συμφωνώ μαζί σας ότι αυτό που είναι ουσιώδες και για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο, είναι να ξαναστήσουμε τον χρηματοοικονομικό κλάδο στα πόδια του για να μπορεί να δανείσει ξανά. Αυτός, αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητά μας. Και εμείς όλες οι αρχές προσπαθούμε να δουλέψουμε στον τομέα αυτό. Τώρα, δεν θέλω να μπω στην, σε κρίση για συγκεκριμένη χώρα, γιατί έχουμε ε, την ευθύνη για 16 χώρες και 329 εκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά σε μια χώρα όπως η δική σας, όπου υπάρχουν πολλά στεγαστικά δάνεια, παρελθόντα δάνεια, πολλά έκρεμη, δηλαδή στεγαστικά δάνεια, που είχαν τιμαριθμοποιηθεί σοβαρά σε σχέση με το 12μηνο Euribor, θα σας πω, αυτή τη στιγμή το Euribor 12 μηνών είναι χαμηλότερο από το LIBOR σε δολάριο για την ίδια διάρκεια και χαμηλότερο από πολλά άλλα επιτόκια της αγοράς και της Τερλίνας ακόμα. Ευχαριστώ. Κύριος Λάγκεν. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στην Επιτροπή μας. Για τις εξηγήσεις σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε με εσάς διάφορα θέματα και ελπίζω να ξανέρχεστε εξίσου συχνά και στο νέο κοινοβούλιο, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμο και για σας και για μας. Έχω δύο ερωτήσεις που σχετίζονται με αυτά που έχουμε ακούσει, αλλά πάνε και λίγο παραπέρα. Ξέρετε, μία συζήτηση που έχει ξεκινήσει σχετικά για το νέο διεθνές αποθεματικό όσον αφορά το σε σχέση με το δολάριο. Ποια είναι η γνώμη σας για την πρόταση αυτή. Είναι ρεαλιστική. Θεωρείτε ότι η πρόταση αυτή έγινε έτσι στην τύχη ή αντικατοπίζει καλύτερα τη νέα διεθνή πραγματικότητα. Και μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με αυτό που είπε και ο κύριος Γκοζές. Όταν συζητιέται το θέμα της χρέωσης στο G20, είναι δυνατόν να προβλεφθεί ένας πληθωρισμός για τα επόμενα τρία χρόνια σε λιγότερο από 2%. Έπειτα, τι γίνεται από τη μεριά των πολιτιών; υπάρχει κίνδυνος πληθωρισμού. Ποια είναι η γνώμη σας. Thank you very much indeed. On the... Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη ερώτηση. Δεν θα σας παραξενέψω αν εξακολουθήσω να αναφέρομαι στην συμφωνηθήσα δήλωση των G7, την οποία εγώ υπέγραψα για το πάρα πολύ αυτό σημαντικό θέμα και που λέει ότι επιβεβαιώνουμε το κοινό μας ενδιαφέρον σε ένα ισχυρό διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα όπου να μην υπάρχει μεγάλη μεταβλητότητα γιατί αυτό θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάκαμψη και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Εμένως αυτό. Αυτό το υπέγραψαν οι επικεφαλής των τραπεζών, ο φίλος μου, Μπερνάνκι και άλλοι ε, διοικητές τραπεζών που πήραν μέρος στη συνάντηση αυτή. Και σημειώνω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επί τη ευκαιρία της τελευταίας ο Τιμ Γκάγκνερ επίση είπε ένα ισχυρό δολάριο είναι προ το συμφέρον της Αμερικανικής οικονομίας. Και ο πρόεδρος Ομπάμα είπε ότι το δολάριο είναι ιδιαίτερα ισχυρό σήμερα και δεν υπάρχει ανάγκη να έχουμε ένα άλλο παγκόσμιο νόμισμα. Σε αυτή τη φάση αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική δήλωση. Δεν προβλέπω τίποτα άλλο στη σημερινή συγκυρία, η οποία είναι πολύ απαιτητική και πολύ ευαίσθητη. Η δεύτερη ερώτησή σας τώρα. Μια γενική παρατήρηση που ισχύει για την νομισματική πολιτική, για τη δημοσιονομική ε, πολιτική, αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε αρχή τώρα που μιλάμε, είναι ταυτόχρονα να είναι τολμηρό ως άμεση απάντηση σε μια κατάσταση η οποία είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Και πιστεύω ότι κι εμείς υπήρξαμε τολμηροί. Λίγες μέρες αμέσως μετά τις αποφάσεις μας σας είπα τι αποφασίσαμε. Αν θυμόσαστε τον Αύγουστο του 2007 ήταν η αρχή η αρχή, η απαρχή μιας θυελώδους φάσης. Ταυτόχρονα αυτό ισχύει και για τις κεντρικές τράπεζες και για τις κυβερνήσεις. Είναι η διάδοση σημασίας να μπορούμε με σαφήνεια να αποδείξουμε την αξιοπιστία μιας στρατηγικής εξόδου από την κρίση. Δηλαδή να δείξουμε ότι ταυτόχρονα είμαστε αποφασισμένοι όλοι να έχουμε μια, ένα βιώσιμη κίνηση προς την ανάκαμψη και μπορούμε να διασφαλίσουμε τους συμπολίτε μας και κατανοώ την ερώτησή σας ότι εμπνέεται δηλαδή ακριβώς από αυτό το μέλημα, να τους διαβεβαιώσουμε λοιπόν ότι μπορεί να υπολογίζουν σε εμά ότι θα τους δώσουμε και τα δύο πράγματα αυτά ταυτόχρονα, σταθερότητα τιμών και ε, δημοσιονομική σταθερότητα. Διαφορετικά θα κάναμε πράγματα που δεν βελτιώνουν την εμπιστοσύνη θα ρίχναμε μπούμεραγκ. Διότι οι συμπολίτε μα είναι έξυπνοι. Και αν δούνε ότι στρώνουμε το δρόμο για ένα αβέβαιο και επικίνδυνο μέλλον, δεν θα έχουν εμπιστοσύνη. Το ίδιο ισχύει για τους επιχειρηματίες, για όλους οι οποίοι συμμετέχουν στις τόσο σημαντικές σήμερα αποφάσεις που θα μας επιτρέψουν πρώτον να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και δεύτερον να επανακινήσει η οικονομία ομαλά, να αποκατασταθεί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να κατανοούμε απόλυτα ότι και οι δύο αυτοί όροι είναι εξίσου σημαντικοί. Κύριε για τους σοσιαλιστές. 1,5 λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ θέλω, όπως και οι άλλοι, να ευχαριστήσω τον κύριο Τρισέ για την συχνή παρουσία του στην Επιτροπή. σε ρωτήσεις και ένα σχόλιο έχω. Για το σχόλιο θα σταθώ σε αυτά που είπατε στις 23 του μηνός στη Wall Street Journal. Είπατε ότι χρειάζεται να ενισχυθούν τα κίνητρα προς την ευρωπαϊκή οικονομία. Εγώ, παρά το ότι κίνητρα. Και αυτό παρά το ότι τα κίνητρα στην Ευρώπη είναι ελάχιστα σε σχέση με το πρόγραμμα ανάκαμψης. Πολύ μικρότερο, για παράδειγμα, από ό,τι κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Τρεις ερωτήσεις τώρα. Ποιος είναι ο στόχος της τράπεζας για την ανάκαμψη. Πότε πιστεύετε ότι θα υπάρξει οικονομική ανάκαμψη όταν αρχίσουν να λειτουργούν οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όταν αρχίσει να ανακάμπτει η οικονομία ή όταν αρχίσει να ανακάμπτει ε, η απασχόληση. Ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεύτερον, θα έπρεπε να εξετάσουμε μία αναζωογόνηση των ε, πιστοτικών αγορών και της τράκια των τραπεζών ενώ δεν έχει ανακάμψει η οικονομία. Δηλαδή, αν οι προοπτικές για τις επιχειρήσεις ε, συνεχίζουν να είναι καταστροφικές, θα, ή, θα παραχωρηθεί, θα παραχωρηθούν περισσότερα δάνεια για την ανάκαμψη της οικονομίας. Και τρίτον, θα ήθελα να ξέρω, ποια πιστεύετε ότι θα υπάρξει ανάπτυξη το 2010. Πιστεύετε ότι θα έχει ολοκληρωθεί η κρίση. Αν όχι, θα χρειαστεί περαιτέρω πολιτική κινήτρων. Γιατί έγιναν τα λάθη που έγιναν. Κύριε Πρόεδρε. Thank you much indeed. Σας ευχαριστώ κύριε μου. Πρώτη ερώτησή σας. Όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο. Να εξασφαλίσουμε ανάπτυξη και δουλειές είναι σαφές. Αλλά το ερώτημα είναι τι κάνει κανείς ακριβώς ενώπιον μιας καταστάσεως όπου έχουν ήδη συσσωρευτεί πολλές ανισορροπίες και όπου γίνεται μια τεραστιά διαστάσεων διόρθωση σε όλες τις αγορές, στην πραγματική οικονομία, σε όλο τον κόσμο. Τι κάνει κανείς λοιπόν ώστε να είναι όσο γίνεται πιο αποτελεσματικός και ε, αποδοτικός για να επιτύχει τον στόχο. Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο να πραγματικά να πούμε δηλαδή ότι κάνουμε λιγότερα από τούτην εδώ την, την ακτή του Ατλαντικού από ότι από την άλλη. Γιατί υπάρχουν του αυτόματου σταθεροποιητέ που είναι πολύ πιο σημαντικοί λόγω ε, των βάσεων του δικού μα συστήματο. Έχουμε μάλιστα και ποσοστά του ΑΕΠ δαπανών που είναι πολύ ψηλότερα στην Ευρώπη από αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά λοιπόν συνδιαμορφώνουν μια κατάσταση και πρέπει κανείς να τα λάβει όλα υπόψη όταν κρίνει. Επίσης, η λήψη υπόψη του παρόντος επίπεδου των ε, αγορών για τα Υπουργεία Οικονομικών, όταν βλέπουμε δηλαδή την κατάσταση εάν οι συμπολίτες μας έχουν εμπιστοσύνη στην βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών μεσοπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα νομίζω όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη λένε ότι κάναν ό,τι ήταν δυνατό επί του παρόντος για να ε, μπορέσουν να επαναχρηματοδοτήσουν το ίδιο χρέος και αυτό που θα έλεγα το γεγονός ότι δηλαδή πρέπει να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών να τους εξηγήσετε ότι πρέπει ε, να μπορούν να, ε, ε, να αντιληφθούν ότι μπορούν να βασίζονται σε εσά. Εμείς πάντως συμφωνούμε με την ανάλυση αυτή. Να πούμε δηλαδή ότι αυτό που κάνουμε πραγματικά τα αποκρίνονται στα αβέλτιστα. Τώρα δεύτερο, πώς θα δανείζει η τράπεζα. Εγώ θεωρώ ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι να υλοποιηθούν αυτά που έχουν αποφασιστεί. Πολλά έχουν αποφασιστεί και πρέπει να υλοποιηθούν. Για τις δύο πρώτες ερωτήσεις η βασική λέξη είναι εφαρμογή. Εφαρμογή, εκτέλεση των αποφασισμένων. Διότι πολλά πράγματα έχουν αποφασιστεί και πρέπει τώρα να τα υλοποιήσουμε. Και αυτό ισχύει και για ε, τις ε, δημόσιες δαπάνες. Επιτάχυνση των δημοσίων δαπανών στη βάση των ήδη ληφθησών αποφάσεων και να γίνουν πραγματικά γρήγορα αυτά που ε, πρέπει. Αυτά που πρέπει σε, είναι απαραίτητο αυτό μέσα σε καταστάσεις όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε τώρα για την Κεντρική Τράπεζα. Εμείς δημοσιεύουμε τώρα τις ε, προγνώσεις μας όπως, βλέπετε, όπως γνωρίζετε δηλαδή ε, τακτικά. Όταν συγκρίνουμε τις δημόσιες προβλέψεις, τις ιδιωτικές προβλέψεις διεθνών οργάτων, ΔΝΤ, ΤΑΦ, Παγκόσμια Τράπεζα κλπ. Βλέπω ότι όλοι μας αναθεωρούμε τις προβλέψεις μας και λαμβάνουμε υπόψη τα νέα δεδομένα, τα νέα νούμερα και δίνουμε φάσμα μεταξύ δύο αριθμών για να δείξουμε ότι παραμένουμε σε έναν κόσμο αβεβαιότητας. Πολλά θα εξαρτηθούν από την ικανότητά μας να επανενέσουμε, να επανεσάγουμε εμπιστοσύνη σε όλους τους φορείς. Καταρχήν στα νοικοκυριά και μετά στις επιχειρήσεις. Εξαρτάται από μας. Αν είμαστε αποτελεσματικοί, αποδοτικοί στο να εφαρμόσουμε αυτά που έχουν ήδη αποφασιστεί, μπορούμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη. Και η οικονομική ανάπτυξη του 2010 θα εξαρτηθεί από εμά. Δεν ε, είναι ο απομηχανής Θεός που θα το αποφασίσει αυτό. Εμείς, η δική μας οικονομική ανάπτυξη εξαρτάται από την ικανότητά μας να επανεισάγουμε εμπιστοσύνη. Η κυρία Βαντεμπούργκ. Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο είναι κατάσταση στα, όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα. Αναφερθήκατε ότι έχει σχέση με τις πληθωριστικές προσδοκίες. Μετά την πρώτη φάση ύφεση, ίσως να υπάρξει ένας υψηλός κίνδυνος πληθωρισμού. Επίσης, ε, υπάρχει συζήτηση να υπάρξουν ομόλογα που να συνδέονται με τον πληθωρισμό τιμαριθμοποιημένα κατά κάποιο τρόπο. Το δεύτερο είναι τα ε, ομόλογα των ε, επιχειρήσεων. Υπάρχει μια πρόταση η τράπεζά σας να παίξει ε, διευθυντικό ρόλο στην έκδοση, όχι στην έκδοση, στην αγορά εταιρικών ομολόγων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μια αγορά που αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Σα ερωτώ λοιπόν ποια είναι η γνώμη σα γι' αυτό. Και ένα τελευταίο σχόλιο, επειδή είναι η τελευταία φορά που εγώ τουλάχιστον πέρα μέρο σε αυτό το διάλογο, θα ήθελα να σα πω κάτι που βγαίνει την καρδιά μου. Προς εσάς, ω επικεφαλή μιας πολυεθνική εταιρεία, κατά κάποιο τρόπο, μεταφέρω λοιπόν αυτή τη φωνή για το τι πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Ίσως υπήρξε κάποια βελτίωση στον κοινωνικό διάλογο και πώς η πληροφόρηση και οι διαβουλεύσεις γίνονται μέσα στην κεντρική τράπεζα. Ελπίζω να καταβάλλετε τις μέγιστες δυνατές προσπάθειες εκ μέρους σας προκειμένου να δώσετε κατά κάποιο ένα μοντέλο λειτουργίας και για τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις και μιλάω και ο του συναδέλφου Μπούλμαν, ο οποίος δεν είναι παρόν, αλλά μου πρότεινε να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Ε, <clears throat> I take good note, of course. Τα σημειώνω βεβαίως. Τα ε, σημείωσα τα τρία σχόλιά σας. Τώρα, για την πρώτη σας ερώτηση είναι σαφές ότι θα περιληφθούν ε, στα ομόλογα και τα, και τα πραγματικά επιτόκια και όπως θα εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια. Και γι' αυτό ο αναμενόμενος πληθωρισμός ε, και ο χειρισμός του θα παραμείνει ε, σημαντικός και είναι εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε σταθερότητα τιμών και να είναι επομένως ασφαλής οι ε, προβλέψεις για τον πληθωρισμό. Είναι σημαντικό αυτό για όλους μας για να είναι και η ανάκαμψη ταχεία Δεύτερο, τα ομόλογα εταιριών είναι η δεύτερη ερώτησή σας. Θα επαναλάβω αυτά που είπα και την τελευταία φορά που απήντησα σε παρόμοια ερώτηση. Η απάντηση είναι ότι θα δούμε τι θα αποφασίσουμε και πότε, εάν αποφασίσουμε κάτι. Τρίτη ερώτηση. την θεωρώ πολύ σημαντική. Θα πω μόνο ότι μετά από πραγματική μελέτη από πλευράς του Εκτελεστικού Συμβουλίου έχουμε πλέον και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνδικάτο και όχι μόνο την Επιτροπή Προσωπικού και αυτό αποδεικνύει ότι θεωρούμε σημαντικό τον κοινωνικό διάλογο. Προηγουμένως είχαμε Επιτροπή Προσωπικού, δεν είχαμε όμως συνδικάτο. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων ο κύριος Κλίντς. Μεγάλο μπουκέτο και από πλευράς μας για τη συνεργασία μας έως τώρα και θεωρούμε ότι πάντοτε με, μας αντιμετωπίσατε με σεβασμό και φιλικότητα και εμείς άλλωστε δεν σας ε, τηγανίσαμε όπως κάνουν στην Αμερική grill session πρόσφατα ήμασταν στην Αμερική λοιπόν και ακούσαμε στην Βουλή των Αντιπροσώπων ότι μας μέμφονται για το γεγονός ότι τα credit for shops γίνονται εδώ σε κεντρική ε, ε, σε κεντρική συγκεντρωτική θέση, συγκεντρωτικά και ότι αυτό είναι δίθεν προστατευτισμός. Έχετε κάποια άποψη. Σε λίγες μέρες άλλωστε θα συνεδριάσουν οι G20 στο Λονδίνο και μου φαίνεται ότι χωρίς να έχει συζητηθεί πολύ στην κοινή γνώμη, υπάρχει μια διαφορετική ερμηνεία των στόχων μεταξύ ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντοτε λέμε ότι όλοι οι τομείς και όλα τα προϊόντα θα πρέπει ε, να ε, τελούν υπορρύθμιση. Ενώ στην Αμερική μας είπαν καθαρά ότι κάθε τομέας που έχει συστημικό χαρακτήρα και σημασία για κάποιο, ε, για σύστημα θα ρυθμιστεί. Πώς το βλέπετε σε αυτό. Το τρίτο αναφέρεται σε κάτι που σας ρώτησε και η κυρία Βαντενμπύρχ. Είπε ο επικεφαλής της ε, Federal Reserve ότι έχει εξαντλήσει πλέον κάθε ε, δυνατότητα που του δίνει το, προστάσιο, το νομισματικό του προστάσιο και το μόνο που μπορεί να κάνει τώρα είναι πλέον να αγοράσει τα τοξικά. Εσείς βλέπετε να έχετε ακόμα κάποιες δυνατότητες. Δεν χρειάζεται να μας πείτε αν θα τις χρησιμοποιήσετε και πότε, αλλά αν καταρχήν βλέπετε ότι διαθέτετε ακόμη κάποιες. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Πρώτη ερώτηση. Για τα credit default swaps. Εμείς θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο ότι έχουμε μια σημαντική βελτίωση στην λειτουργία αυτής της αγοράς. Η κρίση, την κρίση αυτή μοιράζεται και η άλλη πλευρά του Ατλαντικού σε ό,τι μας αφορά ζητούμε ο φορέας που ασχολείται με αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι και εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ο μέγας συνεισφορέας σε αυτήν την μεγάλη αγορά των CDS. Και αυτό σημαίνει πρόοδο για την ώρα. Σε ό,τι αφορά τη διαφορά, την ενδεχόμενη διαφορά απόψεων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει μια σημαντική προσέγγιση και πολύ καλοδεχόμενη μάλιστα. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι καθώς προσεγγίζει η διάσκεψη του G20, η εμπιστοσύνη έχει μεγάλο ρόλο να παίξει, καθώς επίσης η επίδειξη ενότητας και αναμένω και εμείς αλλά και εκείνοι γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική ε, Τράπεζα δεν θα συμμετάσχει στο G20 στο επίπεδο των αρχηγών κατών και διασκέψεων αν και συμμετέχουμε στο επίπεδο των Υπουργών και εγώ θεωρώ ότι η ενότητα απόψεων σε ό,τι αφορά τη διάγνωση και την ανάληψη των απαραίτητων δράσεων η ενότητα σε ό,τι αφορά την ανάγκη αλλαγών, ε, κωδίκων, ε, προτύπων σε σημαντικούς, σε τιματικούς ε, τομείς για την νομισματική σταθερότητα, αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν με σωστό τρόπο. Και νομίζω ότι έχει όντως γίνει μεγάλη πρόοδος, ε, για παράδειγμα και σε οργανισμούς ε, υψηλής μόχλευσης και νομίζω ότι υπάρχει ακόμα και σημαντική συνένεση για παράδειγμα στο 23% του ΑΕΠ, στο 29% του ΑΕΠ από την άλλη μεριά. Και αυτό είναι σημαντικό και ελπίζω <clears throat> ότι η τελική ε, δημοσιονομική δραστηριοποίηση θα φανεί ότι παίζει σημαντικό ρόλο και ότι η ιδέα αυτή ότι η ταχεία εκταμίευση και η ταχεία εφαρμογή των αποφασιστέντων είναι σημαντική και θα μπορέσει όντως να υλοποιηθεί. Αυτά θεωρώ ότι μπορούμε να αναμένουμε από αυτή την ενότητα διάγνωσης αλλά και επίδειξη ενότητας και από τις δύο πλευρές, το Ατλαντικό αλλά και με τον ε, Ειρηνικό και με όλους τους φίλους μας <clears throat> των αναπτυσσομένων οικονομιών. Αφού άλλωστε πρόκειται για παγκόσμια οικονομία, παγκόσμια διάγνωση και παγκόσμια ισχύους αποφάσεις. Εν τέλει, και ίσως μάλιστα να έχω δώσει ήδη το κλειδί για την κατανόηση του ότι πράττουμε από την αρχή της κρίσεως, το 70% της χρηματοδότησης της οικονομίας στην Ευρώπη, στην, στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περνάει από εμπορικές τράπεζες, ενώ στις ΗΠΑ λιγότερο από 30%. Και γι' αυτό εμείς έχουμε ε, επικεντρώσει τα μη στάνταρτ μέτρα μας στην υποστήριξη της ρευστότητας των τραπεζών, με ε, απεριόριστη επιλεξιμότητα για ε, ασφάλιση των τραπεζών και το καθεξής. Και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε και εάν και όταν έρθει ο καιρός θα σας τα πω και με περισσότερες λεπτομέρειες για το τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Πάντως συγκεντρώνουμε τις προσπάθειές μας και σε όλους τους τομείς είμαστε, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω, είμαστε ταχείς στην αντιμετώπιση αυτών των συγκεκριμένων θεμάτων είτε σχετικά με την ε, ε, επιλεξιμότητα των ε, ασφαλιών πρόκειται και για ιδιωτικά χαρτιά με την παροχή απεριόριστης ρευστότητας σε πιο ευρία χρονική βάση για 6 μήνες για παράδειγμα και έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να το κάνουμε αυτό και μέχρι τον επόμενο Ιανουάριο. Ευχαριστώ επανερχόμαστε στην ομάδα του ΕΛΚ, ο Τζον Πέρβης. Ευχαριστώ. Ε, να σας πω επειδή προσωπικά είναι η τελευταία μου, η τελευταία συνάντηση στην οποία συν, συμπαριστάμεθα. Να σας ευχαριστήσω και για την παρουσίαση εδώ και για τον τρόπο με τον οποίο διευθύνεται η Κεντρική Τράπεζα, υποδειγματικού χαρακτήρα θα την έλεγα, και εκτός Ευρωζώνης, εγώ εντυπωσιάστηκα πολύ από τη δουλειά σας. Αναρωτιέμαι ωστόσο, αυτή η ενότητα που επενείται ε, και παγκόσμια και διατραντικά είναι καλή, αλλά μήπως, υπάρχουν μια, μήπως υπάρχει μια κάποια διάσταση απόψεων για τον μεγάλο κίνδυνο. Εσείς λέτε ότι το, ο κίνδυνος είναι ο πληθωρισμός. Πιστεύετε ότι οι εξάδελφοί μας στη ΣΥΠΑ και ίσως και στη Βρετανία φοβούνται τον πληθωρισμό ή τον αποπληθωρισμό. Μήπως ο κίνδυνος της ύφεση ελοχεύει περισσότερο και είναι μεγαλύτερος από τον κίνδυνο του πληθωρισμού. Δεύτερη ερώτηση, βρετανική αν θέλετε. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μέλος της Ευρωζώνης σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Ποιες διαφορές θα υπήρχαν, οι διαφορές μάλλον σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά και τα δημόσια οικονομικά της χώρας θα ήταν πρόβλημα για σας ή θα πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να καθοδηγήσετε τη Βρετανία σε διαφορετική πολιτική, δηλαδή το πρόβλημα δεν θα ήταν δικό σας πια αλλά των Βρετανών. Ευχαριστώ κύριε Πέρβης, για την πρώτη σας ερώτηση. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλες τις παραμέτρους. Την υφιστάμενη κατάσταση, τις τάσεις ύφεσης και αποπληθωρισμού και το ενδεχόμενο αυτές οι τάσεις να γίνουν επεισόδιο, να γίνουν πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν διαφορές εδώ. Οι διαφορές είναι μόνο σε ό,τι αφορά την εκτίμηση που έχει ο καθένας για την οξύτητα του κινδύνου ύφεσης. Ε, αυτή τη στιγμή για τη ζώνη του ευρώ θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κανένας διεθνής οργανισμός, τουλάχιστον όχι εμείς, που θα θεωρούσε ότι ο κίνδυνος ύφεσης είναι υψηλός και τεκμηριωμένος. Βεβαίως πρέπει να επαγρυπνούμε πάντα και αυτό είναι κάτι που, σε το λέω ειλικρινά, πρέπει να το θυμόμαστε. Είμαστε ε, σε εγρήγορση, αλλά τώρα ο κίνδυνος δεν είναι τεκμηριωμένος. Ενώ οι κίνδυνοι πληθωρισμού μέσω πρόθεσμα παραμένουν. Και η διακύμανση από την δημιουργία του ευρώ ήταν πάντα από το 1,7 με 2%. Αυτή είναι η, η διακύμανση των πληθωριστικών των, των αναμον, της αναμονής μας για τον πληθωρισμό μέσω πρόθεσμα. Τώρα, αυτό αν θέλουμε να το δούμε από τον κίνδυνο ύφηση είναι καθησυχαστικό, αλλά πρέπει να είμαστε πάντα ε, στο απίκο. Και δεν πρέπει να μπεδεύουμε μία τάση αποπληθώρησης που οφείλεται στην μείωση των ε, αγαθών και του πετρελαίου και που προκύπτει από την μείωση των, ε, από τη συστολή της Ζήτηση και, και μην ξεχνάτε ότι η αύξηση ε, των τιμών του πετρελαίου ήταν είχε πληθωριστικό χαρακτήρα και οφείλεται στην μείωση της ζήτησης. Το αντίστροφο δεν είναι δεδομένο. Πρέπει να είμαστε πάντα έχοντας καθαρή εικόνα της κατάστασης. Και θα έλεγα ότι έστω κι αν υπήρχε μια ανάλυση του κινδύνου ύφεση διαφορετική και σας το λέω δεν είναι δική μου αρμοδιότητα να χαρακτηρίσω την κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντως εκεί βλέπουν την κατάσταση με διαφορετικό τρόπο, γιατί έχουμε και διαφορετικές καταστάσεις. Ωστόσο όλοι συμφωνούμε ότι μέσο και μάκρο πρόθεσμα ο πληθωρισμός δεν βοηθάει και δεν θα βοηθάει και δεν θα βοηθήσει καθόλου την ανάκαμψη αυτή τη στιγμή. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει ε, σύγκληση, μεγάλη σύγκληση απόψεων στο σημείο αυτό και από τη μία και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και από τη μία και από την άλλη πλευρά της Μάνχης. Δεν θα κάνω πολλά σχόλια για το δεύτερο ερώτημά σας. Νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι είναι προς το συμφέρον της Βρετανίας να είναι μέρος της ζώνης Ευρώπη, πάντα το έλεγα και το λέω. Ξέρω επίσης ότι δεν είναι η άποψη της πλειοψηφίας του λαού του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, είμαι σίγουρος ότι όταν κάποια στιγμή θα το θεωρήσουν ως συμφέρον τους. Ένα πράγμα πρέπει να ξέρετε. Είστε πρόσδεκτοι, αυτό είναι σαφές. Ο κύριος Γκίνερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας συγχαρώ για την ε, στεναρή στάση που πήρε τόσο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας. Θα ήθελα να σα κάνω και εγώ μια ερώτηση για ένα θέμα που ήδη αναφέρθηκε. Τι συμβαίνει στην ευρωπαϊκή οικονομία όπου έχουμε όλο και περισσότερο δαπάνη να χρηματοδοτείται μέσω δημοσίων δανείων. Αναφέρθηκαν χώρες Τώρα φράγει, συνάδελφοι, τι επίπτωση θα έχει αυτό η συνεχής αύξηση της δημόσιας δαπάνης και μέσω εγκυμάτων του προπολογισμού. Το λέω αυτό γιατί μια λύση θα ήταν να έχουμε επιτάχυνση των δημόσιων δαπανών δηλαδή να βγούμε από την κρίση. Και ταυτόχρονα είναι μια τάση που ξεχνάμε ότι δηλαδή οι πληθωριστικές πιέσεις θα υπάρξουν όχι βέβαια μέσα σε ένα μήνα ή σε μία εβδομάδα. Υπάρχει κίνδυνος όμως να επέλθουν όταν θα βρισκόμαστε στην αναδική φάση του κύκλου. Θα ήθελα για παιδαγωγικούς λόγους, αλλά και για πολιτικούς λόγους, να το σχολιάσετε αυτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρος Τρισέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Πιστεύω απόλυτα ότι πρέπει να κάνουμε και αυτό που επιβάλλεται να κάνουμε σήμερα για να αντιμετωπιστεί πολύ δύσκολη κατάσταση σήμερα και να μην ξεχνάμε ότι αν μας διαφύγει ο μέσο μακροπρόθεσμος ορίζοντας βιώσιμης ανάπτυξης, τότε δεν κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε σήμερα, δηλαδή να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη και να επιτρέψουμε στην οικονομία να ανακάμψει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ του βραχυπρόθεσμου και του μέσο μακροπρόθεσμου στοιχείου παραμέτρου στη δημοσιονομική πολιτική. Και τα δύο είναι σημαντικά. Και αν έχουμε και τα δύο, τότε μόνο θα πετύχουμε το στόχο μας. Αν επικεντρώσουμε την προσοχή μας μόνο στα βραχυπρόθεσμα, χάνουμε τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη και τη χάνουμε την εμπιστοσύνη των χρηματαγορών. Και μέσα από αυτά τα δύο κανάλια δεν θα κερδίσουμε, θα χάσουμε. Αυτό είναι το σημαντικό, εμπιστοσύνη σήμερα. Και υπάρχει μία, ένας μόνο ορισμός εμπιστοσύνης. Εμπιστοσύνη για τα νοικοκυριά, για τους επιχειρηματίες, για τις, αγοράς, για τις αγορές εξαρτώνται από αυτά τα δύο. Το τι κάνουμε σήμερα και τι αξιόπιστα δείχνουμε ότι είμαστε σε θέση να κάνουμε μέσω μακροπρόθεσμα και προς το συμφέρον των παιδιών μας. Υπάρχουν ένα σωρό λοιπόν επιχειρήματα για το ότι λειτουργούμε στο optimum. Και το optimum είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη. Κύριε Έτμαρκ, είστε ικανοποιημένο με την απάντηση ή θέλετε να επανέλθετε. Ναι, με ικανοποιεί η απάντηση. Καλό θα ήταν όμως αυτό να ήταν τμήμα της ε, ευρωπαϊκής δημόσιας συζήτησης περισσότερο γιατί το να μην παρεμβαίνει η Κεντρική Τράπεζα στην πολιτική συζήτηση είναι αξιοσέβαστο, αλλά θέλουμε να έχουμε ισορροπία μεταξύ τη νομισματική πολιτική από μια και την άποψη για τη δημοσιονομική πολιτική αφετέρου. Και δεν συζητιέται αρκετά το θέμα αυτό. Ότι υπάρχει μια λύση με αύξηση των δημοσίων δαπανών, αλλά μπορεί ταυτόχρονα να το χάσουμε μέσω νομισματικών επεκτατικών πολιτικών. Είναι λίγο ασύμετρη αυτή η συζήτηση. Σε αυτή τη συζήτηση αναφέρθηκα λοιπόν να μην βλέπουμε μόνο την νομισματική πολιτική αλλά και τη μακροοικονομική προοπτική. Πάντως επαναλαμβάνω η απάντηση με ικανοποίησε. Πρόεδρος Τρισέ, θα ήθελα μόνο να προσθέσω ότι μπορώ να σας στείλω δημόσιες δηλώσεις που έκανα σε μέσα ενημέρωσης και στην Ευρώπη και διεθνώς και λέω όχι περισσότερο για την δαπάνη μέσω προπολογισμού. Είμαστε ήδη στο ύψιστο επίπεδο που θα μπορούσαμε να φανταστούμε και έχει αποδειχθεί και από το κανάλι ισοδυναμιών του Ρικάρντο για να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα των οικονομολόγων και την διαφορά επιτοκίων spreads που παρατηρώ, που παρατηρούμε σε όλες τις αγορές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να σας ε, συγχαρώ. μαζί με όλους αυτούς που επένεσαν την δραστηριότητά σας. Ο κύριος Μπέξελ. Εμείς είμαστε ακόμα εκτός της Ευρωζώνης και πιστεύω ότι θα μείνουμε αρκετά ακόμα εκτός. Μιλάω πάντα για τη χώρα μου. δεν συζητήσαμε πολύ σήμερα για την διεύρυνση της Ευρωζώνης προκειμένου να βοηθηθούν οι χώρες αυτές να εξασφαλίσουν μια σταθερότητα, μια ισορροπία και η σύγκληση ε, να γίνεται σε μακροπρόθεσμη βάση. Αλλά πρόκειται εδώ για έναν ε, φαύλο κύκλο. Από τις χώρες αυτές δημιουργείται κέρδος. Υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών. Τα κέρδη φεύγουν το νόμισμα υποτιμάται. Υπάρχει πρόβλημα στις πιστώσεις. Και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει χωρίς τις ε, συμβουλές προκειμένου να μπούμε κάποτε στην Ευρωζώνη. Δεν ξέρω, η Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να μας βοηθήσει με πράξεις swap ή να μην κάνουμε τίποτα. Βλέπετε τη δυνατότητα ο μηχανισμός των ανταλλαγών να μας επέτρεπε να μπούμε στο ERM ή μόνο θα γίνει αυτό σε μία μοναδική στιγμή νιρβάνα. Βλέπετε να υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί μια αξιόπιστη προθεσμία διορία για αυτούς που θέλουν να μπουν στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Thank you very Ευχαριστώ. Όπως είπα, στην ΕΚΤ έχουμε την άποψη ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε τις και να εφαρμόσουμε τις διατάξεις της ως έχουν, διότι θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό η σύγκληση που απαιτείται βάσει των διαφόρων κριτηρίων πρέπει να επιτυγχάνεται προς το συμφέρον των ενδιαφερομένων χωρών και της ίδιας της ζώνης ευρώ. Η ενδεδειγμένη σύγκληση με βάση τη συνθήκη είναι ουσιαστική κατά την άποψή μας. Εάν μπει μια χώρα στη ζώνη ευρώ να είναι επαρκώς έτοιμη από αυτή τη διαδικασία σύγκλησης, όχι εφάπαξ αλλά και μόνιμα, αν δεν είναι καλά προετοιμασμένη θα αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες η χώρα αυτή. Εάν αντίθετα είναι καλά προετοιμασμένη θα συμβάλλει και στην επιτυχιακή της οικονομίας και ολόκληρης της ζώνης ευρώ. Έχουμε την εντύπωση ότι πιστεύουμε βαθιά ότι υπάρχει συμφέρον, κοινό συμφέρον να προετοιμάσουμε πλήρως και επαγγελματικά όλη τη διαδικασία σύγκλησης. Ξεκινήσαμε 11, τώρα είμαστε 16. Δεν χρειάζεται λοιπόν να αποδείξουμε ότι είμαστε ανοιχτοί στη ζώνη ευρώ, εφόσον είμαστε 16 χώρες. Τώρα, είμαστε βέβαιοι ότι προς το συμφέρον όλων μας είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να οργανώνουμε τη σύγκληση όπως το προβλέπει η συνθήκη. Αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου που είναι παρόμοιες με αυτές που έκανα στην εισαγωγή μου ήταν ένα από τα θέματα που ζήτησε να δουλέψουμε, να, να, μου ζήτησε να σχολιάσω η πρόεδρό σας. Και εγώ να θέσω κάποια ερωτήματα. Πρώτον, βλέπουμε, βλέποντας τα συμπεράσματα της έκθεσης Λαροζιέρ, διαπιστώνουμε ότι το τέλειο είναι για το μέλλον. Τώρα πρέπει να δουλέψουμε με τις υφιστάμενες καταστάσεις. Πιστεύετε ότι ε, η προσέγγιση πρέπει να αλλάξει και στην Κομισιόν γιατί ε, η αντιμετώπιση από την Κομισιόν των μακροοικονομικών ε, διαστάσεων δεν είναι πλήρης. Είπατε ότι είναι επίγον να ξαναπάρουν μπρος οι τράπεζες. Μήπως, αυτό οφείλεται, μήπως το ότι δεν ξαναπαίρνουν μπρος οφείλεται στο ότι έχουν πρόβλημα ιδίων πόρων. Και αν θέλουν να δανείσουν θα πρέπει να ανακεφαλαιώσουν, να αποκτήσουν νέο κεφάλαιο. Άρα πρέπει να προσφύγουν στο κράτος το οποίο με τη σειρά του θα μπει σε αποφάσεις για μισθολογική πολιτική, για stock για φορολογικούς παραδείσους κλπ. Οι συνθήκες λοιπόν των σχεδίων ε, ανάκαμψης των τραπεζών είναι σωστά καθορισμένα. Είμαστε σε καλύτερη κατάσταση αν είχαμε ορίσει ευρωπαϊκά τους όρους, τους ευρωπαϊκούς όρους λειτουργίας των προγραμμάτων ανάκαμψης λαμβάνοντα υπόψη τις επενδυτικές στρατηγικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ομοθεσία για το stock option, τις των φορολογικών παραδείσων αυτά και ε, εισαγωγικά. Μετά για τα toxic assets. Βλέπουμε ότι το θέμα έρχεται και πανέρχεται. Δεν θα δουλέψουμε ως ιστορικοί, αλλά αν ξεκινούσαμε αυτού και από την αρχή, τι θα είχαμε κάνει με αυτά τα τοξικά προϊόντα. Είδαμε πώς ρήπαναν το σύστημα τα subprime ε, τώρα γυρίζουμε γύρω-γύρω και διαπιστώνουμε ότι όσο προχωράει η κρίση, τόσο πιο κρίσιμο γίνεται η ανάγκη να ε, αποτιμήσουμε τα τοξικά προϊόντα. Ακούμε τον Στροσκάμ να λένε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να να προσπαθήσουμε να ξαναστήσουμε το, το σύστημα το τραπεζικό για να χρηματοδοτήσει την οικονομία. Υπάρχουν όμως και οι συμπολίτε μας. Αυτό δύσκολο μπορούμε να το εξηγήσουμε στους συμπολίτε μας. Πώς θα έπρεπε να είχαμε δουλέψει και πώς πρέπει να δουλέψουμε για να οδηγήσουμε στην ανάκαμψη της οικονομίας και της απασχόλησης. Ευχαριστώ. Πρώτη παρατήρηση. Η έκθεση Λαροζιέρ νομίζω όντως πήρε την υφιστάμενη κατάσταση και προσπάθησε να είναι όσο πρακτικότερη γίνεται στις προτάσεις της για να μπορέσει αυτή να, ε, να μπορέσουν ε, να, εφαρμοστούν οι προτάσεις δεδομένων των διαφορετικών απόψεων και ευαισθησιών στην Ευρώπη. Και το καλό της έκθεσης αυτής είναι ότι είναι ακριβώς πρακτική, ότι εντόπισε τα σημεία στα οποία μπορεί να υπάρξει πρόοδος αμέσως. Μπορεί να χρειαστεί να πάμε παραπέρα, το λέει άλλωστε και σε κάποια κομμάτια η έκθεση. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Για την Επιτροπή τώρα, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι στις επαφές που είχαμε στην τράπεζα με την Επιτροπή, έχουμε επαφές με πολλούς επιτρόπους, ε, με τον κύριο Αλμούνια κατά βάση, αλλά και με άλλους. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι ευτυχής για, όλες, για όλο το πλαίσιο των σχέσεών μας με την Επιτροπή. Σε κάθε τομέα διαπιστώνω ότι υπάρχει η Επιτροπή είναι, είναι επαγγελματική, έχει ενιαία θέση. Δεν νομίζω να υπάρχουν δυσκολίες που να σχετίζονται με την... τον αριθμό των εμπλεκόμενων επιτρόπων. Τρεις επιτρόπους βλέπω κατά βάση, αλλά διαπιστώνω ότι υπήρχε πολύ καλός βαθμός ενότητας μεταξύ τους και μπορέσαμε να υπερκεράσουμε πολλές δυσκολίες και αυτήν που δεν είναι απλή για την Επιτροπή να πρέπει να εξασφαλίσουμε ισότιμη ε, ισότιμο ανταγωνισμό στην Ευρώπη, καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, εν, επιτρέποντας ταυτόχρονα στα κράτη να κινητοποιηθούν για να ε, βοηθήσουν το ταραγμένο δικό τους χρηματοοικονομικό σύστημα. Δεύτερη ερώτηση. η Επιτροπή χρειάστηκε να αντιμετωπίσει ένα μείζον ζήτημα. Η Κεντρική Τραπεζα είπε στα κράτη υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα φράγμα έναντι του κινδύνου συστημικής έλψης συστημικής έλλειψης ρευστότητας. Αλλά εμείς ως τράπεζα δεν έχουμε την ε, δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα φράγμα για την συστημική αφαιρεγκαιότητα και η Επιτροπή γρήγορα και σε πολύ δύσκολες συνθήκες χρειάστηκε να προετοιμάσει ένα τέτοιο σχέδιο. Και νομίζω ότι τα κράτη κατάφεραν να λάβουν πολύ σημαντικές αποφάσεις πολύ γρήγορα. Εγώ θα έλεγα ότι η Ευρώπη με, τις θεσμικές, με τη θεσμική πολυμορφία της, δεν είμαστε πολιτική ομοσπονδία ολοκληρωμένοι, δεν υπάρχει ένα κεντρικό σημείο λήψη αποφάσεων όπω στι ΗΠΑ. Ωστόσο, παρά τα αυτά, οι ενδεδειγμένε αποφάσει λήφθηκαν. Μπορούμε να πούμε, θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει καλύτερη δουλειά ε, ή πολύ καλύτερη δουλειά, αλλά δεν υπάρχει στην Ευρώπη το αντίστοιχο των Lehman Brothers, ούτε το μείζον πολιτικό πρόβλημα που εμφανίστηκε αλλού για την αποδοχή ή όχι ενός φιλόδοξου προγράμματος καταπολέμησης της συστημικής αστάθειας. Ωστόσο και οι αποφάσεις λήφθηκαν από τα κράτη, από τις κυβερνήσεις και από την ε, Επιτροπή. Τρίτη ερώτηση. Τα τοξικά προϊόντα, τα toxic assets. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Κανείς δεν είναι πάνσοφος. Η κατάσταση εξελίσσεται συνεχώς. Δεν νομίζω λοιπόν ότι εκπλήσει πως αυτή τη στιγμή έχουμε τρεις μεγάλες εναλλακτικές επιλογές. Ανακεφαλαιοποίηση, εγγύησεις για την μέσο και μακροπρο αναχρηματοδότηση των τραπεζών και ένα τελευταίο πιο πρόσφατο στοιχείο για μας στην Ευρώπη και που επανεργοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες η αντιμετώπιση με διαφορετικά μέτρα των τοξικών προϊόντων. Δεν με εκπλήσει το ότι εδώ βρισκόμαστε και έχουμε αυτή την επιλογή η Σοσιαλιστική Ομάδα, στην Φερέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους συναδέλφων που είναι απόντες θα μιλήσω. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ζώντας μια κρίση, έχουμε και την ευκαιρία να δούμε πιο ουσιώδη θέματα, παρότι όταν τα πράγματα είναι business as usual. Δηλαδή, ήθελα την άποψή σας αν συζητήσετε το θέμα της βιωσιμότητας του κοινού νομίσματος, τη στιγμή που έχουμε τόσο ασύμετρες δράσεις μεταξύ των χωρών και μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούν το ευρώ και μεταξύ αυτών που βρίσκονται εκτός ευρώ. Είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα αυτό, διότι ακόμα και αν καταφέρουμε να κρατήσουμε το ευρώ, αυτό δημιουργεί σοβαρά πολιτικά προβλήματα. Έπειτα αυτές οι ασύμετρες επιδράσεις διευρύθηκαν με την κρίση και τα μέσα αντίδρασης είναι τελείως διαφορετικά σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Το συζητάτε το θέμα αυτό. Ποιες είναι οι απόψεις Είναι βιώσιμο σε αυτή τη φάση που ζούμε. Ευχαριστώ. Απάντηση. Έχουμε δύο ερωτήματα διαφορετικά εδώ. Το ένα ερώτημα είναι για την ίδια την Ευρωζώνη. Και ε, το άλλο ερώτημα είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωζώνη αφενό και άλλες χώρες με διαφορετικά νομίσματα αφετέρου. Για την Ευρωζώνη. Ξέρετε ότι αναλύσαμε αρκετά τις διαφορές και τις ομοιότητες. Σε μια μεγάλη υπηρετική οικονομία όπως είναι η Ευρωζώνη και μια άλλη ζώνη όπως είναι οι Ηνωμένε Πολιτείες. Και είχα την ευκαιρία ήδη να σας εξηγήσω και στο παρελθόν ότι βρίσκουμε την ίδια τάξη μεγέθους στάνταρ απόκλησης για τον πληθωρισμό, για την οικονομική ανάπτυξη. Τον ίδιο φάσμα διασποράς όσον αφορά την, το παραγωγή κατά, κατά μονάδα εργασίας. Η υπογραφή της Καλιφόρνιας δεν είναι ίδια με την υπογραφή του Wyoming ή το, της Μασάχουσέτης. Έχουμε και εκεί διαφορές, έχουμε και εδώ διαφορές, αλλά και στις δύο περιπτώσεις έχουμε κράτη και χώρες που βρίσκονται σε διαφορετική κατάσταση. Και είναι σωστό αυτό, διότι υπάρχουν στην κάθε περιοχή ειδικά χαρακτηριστικά, όπως και εσείς είπατε. Όλα τα σοκ δεν είναι συμμετρικά. Ωστόσο, όσον αφορά την ίδια τη φύση των σοκ και των δονήσεων και στην Ευρώπη και στην Αμερική, πολλοί οικονομολόγοι λένε ότι υπάρχει περισσότερη συμμετρία στη δική μας περίπτωση, διότι οι οικονομίες των κρατών μας, των κρατών εθνών της Ένωσης είναι πιο διαφοροποιημένες από ότι οι πολιτείες στις ΗΠΑ που είναι κάπως πιο εξειδικευμένες, γιατί εκεί βρίσκονται σε μια ενιαία αγορά με ένα ενιαίο νόμισμα εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό. Επαναλαμβάνω, στην Ένωση έχουμε μια ενιαία νομισματική πολιτική, την έχουμε αριστοποιήσει στο επίπεδο αυτών των 329 εκατομμυρίων ανθρώπων που ανάφερα και όλα το υπόλοιπο πλωστάσιο που διαθέτουν οι κυβερνήσεις και οι κοινωνικοί εταίροι προκειμένου να προσαρμοστούν στην συγκεκριμένη κατάσταση κάθε φορά που και χρονικά μερικές φορές είναι πολύ επίγουσα και απαιτητική και σε κάποια άλλη φάση λιγότερο απαιτητική. Σήμερα φυσικά η κατάσταση είναι απολύτως απαιτητική για όλους τους εταίρους, όχι μόνο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παγκόσμια. Και μετά έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο, ως σύνολο, με διαφορετικές καταστάσεις και εδώ. Το είπα και στην εισαγωγή μου και μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των εθνών. Μερικοί έχουν ένα βαθμό ευελιξίας, ελαστικότητας αξιοθαύμαστο και δεν είναι περίεργο αυτό, εξηγείται. Για διάφορους λόγους έχουν καλύτερες μακροπολιτικές από ότι άλλες χώρες που έχουν δυσκολίες. Και ήδη μερικές έχουν βοηθηθεί και από την Κομισιόν και από την Ένωση και από το ΔΕΛΤΑ πρέπει να αναγνωρίσουμε τις διαφορετικές καταστάσεις και να μην έχουμε την ίδια μέθοδο παραδείγματος χάρη για τις κέντρο-ανατολικές χώρες μέλη της Ένωσης σαν ήταν μια ενιαία οντότητα. Και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές. Οι χώρες ίδιες το τονίζουν αυτό, ότι είμαστε διαφορετικές λένε και το, το πιστεύω ότι είναι διαφορετικές. Πρέπει να προσαρμοστούμε και εμείς και η Ένωση και η Κομισιόν και το Συμβούλιο και προσαρμόστηκαν προκειμένου να λάβουν υπόψη αυτές τις διαφορετικές καταστάσεις. Κύριε Σας ευχαριστώ. Με τη σειρά μου ευχαριστώ τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και τον συγχαίρω για την σοφροσύνη του που σίγουρα έχει συμβάλει στην ευημερία πολλών Ευρωπαίων. Επανέρχομαι στο θέμα των μη ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως μη, χωρών, ε, των χωρών που δεν εντάσσονται στη ζώνη ευρώ, κυρίως ε, κεντρικών και ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών. Σας παρακαλώ κύριε μου κόβετε τη θέα. Ωστόσο υπάρχουν λόγοι που συνηγορούν υπέρ μιας επιτάχυνσης της ένταξης που ίσως είναι το λιγότερο από τα δύο προκείμενα κακά. Είναι καλύτερα να υπάρχει μία σταθερή, ένα σταθερός χώρος ε, στην Ευρώπη. Ωστόσο ορισμένες φορές ε, φοβούμε ότι έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί ορισμένες χώρες που έχουν μπει στη ζώνη ευρώ και που ήδη ήταν πολύ απομακρυσμένες από τα πρότυπα και τα επίπεδα όταν εντάχθηκαν και στην ουσία ποτέ δεν τα, δεν τα κριτήρια αυτά και τώρα κατευθύνονται στην, προς την άλλη κατεύθυνση. Πώς επιτρέπεται να είμαστε τότε υπεραυστηροί σε ό,τι αφορά την πλήρωση των κριτηρίων ένταξης από τις χώρες για τις οποίες ομιλούμε. Και ίσως πρέπει να υποστηρίξουμε μέτρα υπέρ των χωρών αυτών που έτσι κι αλλιώς η ένταξή τους δεν πρόκειται να επηρεάσει κατά πολύ την πορεία της ζώνης ευρώ. Μήπως μπορούμε να αποδειχθούμε ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ. Κατανοώ την ερώτησή σας. Κατανοώ γιατί κάνετε τα σχόλια αυτά. Θα συνεχίσω να ισχυρίζομαι ότι προς χάρη των ίδιων των χωρών αυτών που αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις ορισμένες από αυτές. Πάλι νομίζω ότι θα ήταν πρόωρο να θεωρήσουμε ότι η λύση είναι να ενταχθούν στη ζώνη ευρώ ακόμη και αν δεν είναι απόλυτα προετοιμασμένες. Γιατί αυτό σημαίνει σιωπηρά αυτή η ιδέα της επιτάχυνσης της ένταξης που σημαίνει δηλαδή ότι θα ενταχθούν χωρίς να πληρούν πλήρως τα κριτήρια. Ήδη μη, αν ε, δεν ισχύει αυτό δεν υπάρχει επιτάχυνση. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διατηρήσει την θέση αυτή ότι θέλουμε να ισχύει ολόκληρο το περιεχόμενο της συνθήκης και όλης της συνθήκης σε όλη αυτή την πορεία μέχρι την ένταξη που βεβαίως δεν είναι κλειστό χώρο, δεν είναι κλειστή λέσχη. Από 11 περάσαμε σε 16 και θα συνεχίσουμε να διευρυνόμαστε πάντοτε με βάση τη συνθήκη. Πρέπει να διατηρήσουμε νομίζω τους κανόνες αυτούς που είναι άλλωστε προς το συμφέρον όλων. Η ιδέα ότι δήθεν επειδή βρισκόμαστε σε κρίση πρέπει να επιταχύνουμε την ένταξη στην ζώνη ευρώ ορισμένων χωρών νομίζω ότι δεν εντάσσεται δεν συμβαδίζει με την ιδέα ότι η ένταξη στη ζώνη ευρώ σημαίνει κιόλας ότι μοιράζεται μια χώρα, μια κοινή μοίρα για ένα πολύ πολύ μακρό χρονικό διάστημα, μια κοινή, ένα, ένα κοινό πεπρωμένο. Δεν είναι απλώς για να αποφευθούν κάποιες δυσκολίες από εδώ και από εκεί τώρα, είναι βεβαίως όπως είπα να ε, ενταχθούν σε μια ομάδα η οποία θα έχει ένα κοινό μέλλον, μια κοινή μοίρα. Κάποια στιγμή θα γίνουμε 25 οι χώρες του ευρώ, διότι 25 χώρες έχουν το δικαίωμα να μπουν στο ευρώ, στη ζώνη ευρώ, όταν θα ε, πληρούνται τα κριτήρια. Και δύο από τις 27 ε, επιθυμούν να μείνουν εκτός. Όμως από αυτές τις δύο η Δανία έχει ένα opt-out, παρόλα αυτά ακολουθεί τις πολιτικές μας. Υπάρχει χώρος για μια ερώτηση, χρόνος μάλλον για μια ερώτηση από πλευράς Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Για ένα μισή λεπτό η κυρία Λούλινγκ. Σύντομη, πρόεδρε. Μια παράξενη ερώτηση έχω, που δεν καταλαβαίνω. Έμαθα ότι η Κεντρική Τράπεζα του Λουξεμβούργου δάνεισε 800 εκατομμύρια ευρώ στην Κάουπτιν Bank και ένα δις στη Banking. Τι άποψη έχετε. Υπάρχει κάποια συνεννόηση, γιατί ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Ευχαριστώ. La Banque Centrale μου, η Κεντρική Τράπεζα του Λουξεμβούργου είναι μία από τις κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος και εφαρμόζει στο Λουξεμβούργο τους κανόνες του συστήματος όπως η Bundesbank εφαρμόζει τους κανόνες στη Φραγκφούρτη και κάθε κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ εφαρμόζει τους δικούς της κανόνες. Και το Λουξεμβούργο το ίδιο. Μαζί είμαστε η κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ όλοι μαζί και εφαρμόζουμε τους κανόνες εγγυήσεων και επιλεξιμότητας για τη ζώνη ευρώ. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, εσείς είστε καλύτερα ενημερωμένοι από μένα, τώρα τουλάχιστον, αλλά δεν αμφιβάλλω ότι λόγω της θέσης της ως μέλος του συστήματος Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών, η Τράπεζα του Λουξεμβούργου κάνει αυτό που πρέπει και παρέχεται η απαραίτητη υπάρχουν οι απαραίτητες εγγύσεις. Άλλη ερώτηση για το ΕΛΚ. Ο κύριος Πέρβης. Τα περιθώρια δημοσίου χρέους των ζωνών, των χωρών της ζώνης Ευρώπη ε, αυξάνονται, έτσι, διευρύνονται και δικαίως. Υπάρχει ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης των εξαιρετικά υψηλών δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα κράτος μέλος όταν δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος του. Έχετε ένα πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης. Σας ε, αναφέρθηκα στα spread πριν από λίγο όταν είπα ότι Υπάρχει κάποια στιγμή που πρέπει να λάβεις υπόψη τις αγορές όταν σχεδιάζεις τη φορολογική δραστηριοποίησή σου. Κάτι αναγκαίο και στη ζώνη του ευρώ και αλλού στον κόσμο. Εμείς έχουμε μηνύματα που δείχνουν ότι χρειάζεται να είναι κανείς επιφυλακτικός, προσεκτικός και να μην δρά ε, απερίσκεπτα. Δεύτερον, έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις της ζώνης ευρώ ότι θα είναι υπεύθυνε και για τη δική τους αξιοπιστία και για την αξιοπιστία του συστήματος. Το λέω, εμείς εμπιστευόμαστε τις κυβερνήσεις της ζώνης ευρώ ώστε να προστατεύσουν την αξιοπιστία και την πιστοληπτική τους ικανότητα. Κάτι, αυτό είναι αναγκαίο, ξέρετε, στη ζώνη ευρώ κάθε κυβέρνηση, σωστότερα κάθε κοινοβούλιο είναι υπεύθυνοι για την φορολογική πολιτική που ασκούν. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα στον τομέα αυτό και πάλι να σας πω το εξή. Απαντώ σε μια ερώτηση που δεν θέσατε. Αν με ρωτούσατε θα σας έλεγα ότι είναι παράλογο να φαντάζεται κανείς ότι μία χώρα στη ζώνη του ευρώ θα ήταν σε τέτοια κατάσταση που θα δημιουργούσε πρόβλημα για τη ζώνη αυτή καθ' αυτή. Άλλη ερώτηση για τους σοσιαλιστές, κύριε Βαντεμπούλκ. Um, you πολύ κατηγορηματικός λέγοντας ότι υπάρχει προσέγγιση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης. στην προετοιμασία για το G20 για την εποπτεία συστημικών κινδύνων ή των του κλάδου γενικά. Δεν είπατε όμως προς ποια κατεύθυνση γίνεται αυτή η σύγκληση. Μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένος. Απάντηση. Αυτό που είπα και έχετε δίκιο να θέτετε το ερώτημα είναι ότι η προσέγγιση είναι κυρίως προς την κατεύθυνση αποδοχής ότι απαιτείται ένα σωστό επίπεδο ρυθμίσεων και εποπτείας. Η τελευταία δήλωση και του Υπουργού Οικονομικών Γκάιτλερ και από τον Πρόεδρο των Πολιτειών υπήρξε σαφής. Επίσης και η δήλωση του Γκόρντον Μπράουν ήταν αρκετά σαφής. Βλέπουμε μερικές αλλαγές και δεν με παραξενεύει αυτό, γιατί τα γεγονότα είναι μπροστά μας. Τα βλέπουμε όλοι. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν θεωρώ και δεν πρέπει να μας παραξενεύει αυτό, δημιουργείται η αίσθηση ότι για να επιτρέψουμε στην παγκόσμια οικονομία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι περισσότερο ελαστικό, λιγότερο εύθραυστο, να τίνει λιγότερο προς απότομες ανόδους και καθόδους, επιβάλλεται να έχω μια σωστό χειρισμό και μεταχείριση όλων των στοιχείων του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Με βάση όλες τις πληροφορίες που έχω, θεωρώ ότι υπάρχει ευρεία συνένεση ότι χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη διαφάνεια για τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, θεσμικά όργανα και αγορές, πολύ λιγότερο βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα δράση, που ήταν μια τρέχουσα συμπεριφορά, πολύ περισσότερη αποτελεσματική μάχη κατά των ε, στοιχείων που δρούν υπέρ της ανωδική φάσης του κύκλου και όλα αυτά θα, σαν αυτά θα συμβάλλει και τα διάφορα φόρουμ που αναφέρθηκαν οικονομικής σταθερότητας, όλοι οι εταίροι στις μεγάλες αγορές, στο επίπεδο της παγκόσμιας, του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και οι υπουργοί των G20 η και η Γενική Τραπεζίτη, στο οποίο πήρα μέρο, νομίζω εκεί διαπιστώθηκε ευρεία συνένεση. Βέβαια, όταν πάμε να εφαρμόσουμε, και το λέω, η ουσία είναι η εφαρμογή. Γρήγορη, αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων. εκεί να διαπιστώσουμε ότι τα πράγματα είναι κάπως πιο περίπλοκα. Όσον αφορά όμως τη διάγνωση, τους διάβλους λύσεις για, για να γίνει πιο ελαστικό το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, βλέπω ότι υπάρχει συνένεση και στον ε, στις γεωμηχανικά ανεπτυγμένες χώρες και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και όλοι οι οικονομολόγοι με βάση τις τρέχουσες πληροφορίες. Και σε μερικές μέρες ή μισές μέρες θα έχουμε την περίφημη αυτή διάσκεψη των G20. Για τους φιλελεύθερους η κυρία Στάρκεβιτσούτα. Μία ερώτηση ευθεία. Τέτοιες ερωτήσεις ρωτούν συνήθως οι πολίτες. Κύριε Τρισέ, πότε μπορούμε να περιμένουμε την ανάκαμψη της οικονομίας. Βιώσιμα τουλάχιστον. Αυτό είναι το σημαντικότερο ερώτημα των πολιτών. Κατόπιν, μερικές φορές λέγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη για την διεύρυνση γιατί η Ιρλανδία δεν έχει επικυρώσει τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η Ευρωζώνη τι γίνεται. Είναι έτοιμη η Ευρωζώνη για διεύρυνση. Είπατε ότι διευρύνθηκε από τα 11 στα 16 μέλη. Έχετε προβλήματα διαχείρισης νομισματικής πολιτικής Τη Λισαβόνα, μήπω και εσεί χρειάζεστε μια συνθήκη τη Λισαβόνα, μικρού μεγέθους. Ευχαριστώ. Πρώτη ερώτηση. Αυτό που βλέπουμε σήμερα και αυτό λένε και οι εικασίες δημόσιες και ιδιωτικές και δεν απομακρύνουμε από αυτέ τις προβλέψεις και οι δικές μας και των άλλων προς τα ίδια προς τις ίδιες, ε, ίδια, την ίδια κατεύθυνση έχουν έστω και τα νούμερα είναι διαφορετικά λένε όλοι το 2009 είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά με αρνητική αύξηση όλη τη χρονιά. Το 2010 αν κάνουμε ό,τι χρειάζεται, χωρίς λάθη, αν επαναφέρουμε την, αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη που χάθηκε σε διάφορες βασικές δομές, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, θα παγιωθεί η ανάκαμψη στα μέσα κατά τη διάρκεια του 2010. Αλλά αυτό δεν είναι δεδομένο. Από εμά εξαρτάται εάν κάνουμε αυτό που απαιτούν, αυτά που απαιτούν οι πολύ δύσκολες περιστάσεις. Είμαι, πιστεύω ότι θα υπάρχει αυτή η ανάκαψη το 2010. Διεύρυνση της Ένωσης τώρα και της ζώνης του ευρώ. Διαφορετικά θέματα για τη διεύρυνση της Ένωσης είναι αρμοδιότητα άλλων οργάνων, όχι της ΕΚΤ. Για τη ζώνη του ευρώ, να σας επιβεβαιώσω ότι δεν είμαστε κλειστό μαγαζί. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ξεκινούσαμε το ευρώ με 11 χώρες. Δεν το θυμάμαι. Εγώ ήμουνα στι διαπραγματεύσει για τη συνθήκη του Μάαστριχτ και θυμάμαι τι σκεφτόμασταν, ποιες χώρε είχαμε υπόψη για το ξεκίνημα της, του ευρώ. Πολύ λιγότερε από 11. Το ότι 11 ήταν μέλη ήταν τεράστια επιτυχία. Κανεί δεν μπορούσε να φανταστεί ότι 10 χρόνια μετά θα ήμασταν ήδη 16. Πρόκειται για μια διαδικασία ιστορικού χαρακτήρα, τεράστια εμβέλεια και πολύ γρήγορη δεν είμαστε κλειστό μαγαζί. Σας είπα ότι θα διευρύνουμε, θα διευρυνθούμε βάσει τις συνθήκες μέχρι τον αριθμό των 25, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό πρέπει να γίνει με πολύ επαγγελματικό τρόπο. Μιλάμε για πολύ σοβαρά θέματα η κοινή διαχείριση ενός ενιαίου πεπρωμένου. Τούτο πρέπει να γίνει όσο πιο επαγγελματικά γίνεται γιατί είμαστε υπεύθυνοι σήμερα για 329 εκατομμύρια πολίτες που χρησιμοποιούν το νόμισμα αυτό και αύριο θα είμαστε για περισσότερους. Προς το συμφέρον λοιπόν όλων των χωρών και όλων των ομάδων χωρών πρέπει να είμαστε επαγγελματίες και το λέω αυτό έχοντας τη συνείδηση του βάρους της αποστολής μου. Είμαστε με 16 χώρες περισσότεροι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ευθύνες αυτές πρέπει να τις έχουμε υπόψη μας. Θέλετε να επανέλθετε κύριε Στακεβιτσιούτε. Ε, ε, ασφαλώς πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι αλλά έχω την θαυμάσια ομιλία σας του Δουβλίνου και που αναφέρεστε σε τέσσερων, τεσσάρων ειδών χώρες μέσα στην ε, ζώνη ευρώ. Η Λιθουανία, η χώρα μου, ταιριάζει απολύτως στην τέταρτη κατηγορία των χωρών που είναι μέσα στην ζώνη ευρώ. Και εξακολουθώ να να μην καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά. Απάντηση. Ίσως μπορώ να μπω σε θέματα πιο τεχνικού χαρακτήρα. Θα θυμάστε τι έγινε και η απόφαση ελήφθη από το Συμβούλιο Υπουργών μετά από σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με ε, την ε, αξιολόγηση βέβαια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά ε, βεβαίω σημειώνω αυτό που είπατε κυρία μου. Μας μένει λίγος χρόνος κατ' εξαίρεση και υποφελούμε για να επανέλθω σε κάποια σημεία. Όπως ξέρετε συζητούμε τώρα την αναθεώρηση της οδηγίας ε, CRD και συζητούμε με τον με συζητήσαμε με τον κύριο Βίλινγκ το όριο παρακράτησης που πρέπει να επιβάλλεται στις τράπεζες όταν εκδίδουν ε, σύνθετα προϊόντα. Η συζήτηση έγινε ότι λέμε ότι οι Αμερικανοί λένε 10% θα μπορούσαμε Μάλλον εμείς λέμε το 20% θα ήταν ένα εμπόδιο, ένα πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό αυτό. Η άποψη της τράπεζας, πέραν της άποψης της τράπεζας για την οδηγία μπορείτε να μας δώσετε την προσωπική σας άποψη. Δεύτερο ζήτημα. Είπατε στην κυρία Βαντεμπουργκ ότι υπάρχει σύμπνοια με, τους, με τη ΣΥΠΑ ε, στην αντιμετώπιση των τοξικών προϊόντων. Εμείς με τον κύριο Βίλεγγ είχαμε πει και αυτό συμφωνούσε μαζί μας ότι όταν εξετάζουμε τα συμπεράσματα των Υπουργών Οικονομικών του G20 υπάρχει η εισαγωγή της έννοιας της συστημικής ε, οντότητας αυτή η συστημική διάσταση μήπως υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της αρχής ότι κάθε όργανο που δραστηριοποιείται στην χρηματοοικονομική αγορά θα πρέπει να ρυθμίζεται, να εποπτεύεται σε ό,τι αφορά το βαθμό διακινδύνευσης ή ε, χρέους της. Μήπως εν τέλει επαναδημιουργηθεί ένα σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Μιλήσατε μετά για την σημασία των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Πιστεύετε ότι το ποιοτικό άλμα που πρέπει να γίνει μεταξύ των συμπερασμάτων του G20 στην Ουάσιγκτον και του επερχόμενου Εμείς δεν είμαστε ειδικοί, αλλά ποια είναι η άποψη που υπάρχει για αυτές τις ε, μακροοικονομικές παγκόσμιες ανισορροπίες. Ευχαριστώ. Πρώτη ερώτηση. Θα έλεγα. Σε αυτό που σας είπε ο πρόεδρος της ε, Επιτροπής της Βασιλείας είναι πρόεδρος και έχει σημαντική ευθύνη. Να και είναι αρμόδιος να υποβάλει προτάσεις που θα αντιστοιχούν στην ενίσχυση της σταθερότητας και της ανθεκτικότητας των διεθνών οικονομιών και να κάνει το updating των αναγκαίων διατάξεων που μετά από το stress test αυτό σε φυσικό μέγεθος που περνάει ο κόσμος και που δεν εμφανίζεται να είναι αρκετά αντικυκλικό. Η δυσκολία που έχουμε είναι να καταλάβουμε σωστά τι είναι αναγκαίο για να είναι πιο ανθεκτικό το σύστημα. Χρειαζόμαστε τα τελευταία 15 χρόνια μάλλον κατά τα τελευταία 15 χρόνια, για διάφορους λόγους και μετά από πιέσεις και των ίδιων των αγορών, καταργήσαμε μια σειρά ε, προστατευτικών δικλείδων, όπως για παραδείγματος χάρη το dynamic provisioning, το εκ των προτέρων η ε, εκτομετώ αξιολόγηση των ε, στοιχείων του ενεργητικού. Αυτό που κάνανε οι Ισπανοί. Γιατί, γιατί οι φορολογικές ε, υπηρεσίες θεωρούσαν ότι αυτό μείωνε τα έσοδα και άρα ήταν κακό. Βλέπουμε όμως το, τη σημασία του να έχουμε κάποια προστατευτικά μαξιλαράκια. Άλλο θέμα. Ε, ένα αυτοκίνητο. Ε, σαν να είμαστε σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε του κόσμου τα airbag αριστερά-δεξιά και σταδιακά βγάζουμε όλα τα, όλα, τα, τα airbag και ε, γίνεται ένα τύχημα και είμαστε τραυματισμένοι παντού. Πρέπει να δεχθούμε λοιπόν ότι η προηγούμενη περίοδος ήταν μια περίοδος που για διάφορους λόγους, κατανοητούς όλους, ιδιαίτερους, λόγω της συμπεριφορά των εποπτικών αρχών, των λογιστικών υπηρεσιών, των ε, ε υπεύθυνων ελέγχου της χρηματαγοράς, δεν είχε προστατευτικά και Τώρα πρέπει να ξαναδούμε σε παγκόσμιο επίπεδο την σταθερότητα της διεθνούς χρηματοοικονομικής κατάστασης. Για το δεύτερο θέμα, είναι σαφές ότι η προσέγγιση που θεωρώ σημαντική, ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ, ε, υπάρχει. Προφανώς υπάρχουν κάποιες διστάμενες απόψεις, κάποιες πάντων αποκλίνεις απόψεις σε ό,τι αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο και σας λέω ότι δεν ρυθμίζουμε μόνο και μόνο γιατί μας αρέσει να ρυθμίζουμε, αλλά για να είναι ανθεκτικό το σύστημα. Τώρα, συστημική οντότητα δεν με σοκάρει σαν όρος και αυτό περιλαμβάνεται και στο ανακοινωθέν του G20 Το υπέγραψα και εγώ και δεν κάνω πίσω. Αλλά το ότι είμαστε ικανοί να δείξουμε ότι με ενιαίο τρόπο κάνουμε τη διάγνωση και με ενιαίο τρόπο κάνουμε ε, την αναζήτηση των όρων είναι βασικό στοιχείο για την αξιοπιστία μας. Τελευταίο θέμα. Πολύ σημαντικό και δεν το αναφέραμε μέχρι τώρα. Όταν λέμε τι χρειάζεται για να, επιτύχουμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, απαντώ. Ότι χρειαζόμαστε και δεν το λέω με βάση το μέγεθο τη σπουδαιότητα, να υπάρξει υποστήριξη της χρηματοποίηση πιστοτική σφαίρας. Να ξαναρχίσουν τα δάνεια οι τράπεζε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να υλοποιηθούν αυτά που αποφασίστηκαν. Αυτό είναι ήδη σημαντικό. Χρειάζεται η μεταρρύθμιση των ρυθμιστικών δραστηριοτήτων standards and codes, προληπτικός έλεγχος, μεγαλύτερη διαφάνεια, λιγότερη βραχυπρόθεσμη στρατηγική και περισσότερη αντικυκλικότητα στο σύστημα. Όμως ταυτόχρονα χρειάζεται να εποπτεύουμε και να παρακολουθούμε τις μακροοικονομικές πολιτικές. Χρειάζεται σε μια παγκόσμια οικονομία, πραγματικά παγκοσμιοποιημένη τώρα, μια, μια σημαντική παράμετρο, να υπάρχει ένα δούνο του με πραγματική μακροοικονομική δυνατότητα εποπτείας και μια συνένεση των βασικών κρατών ή οικονομικών ενωτήτων όπως η ζώνη του ευρώ, μια επαρκή απόφαση να, να, να, ασκούν πιέσεις στις άλλες κυβερνήσεις. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να συσσωρεύσουμε ανισορροπίες και να ξαναβρεθούμε με ένα σύνολο ε, ανισορροπιών που θα προκαλέσουν μια νέα κρίση. Ο τελευταίος λοιπόν πυλώνας των αναγκών μας είναι, σε εισαγωγικά αυτά, είναι μια συνένεση των κρατών ή των οικονομικών ενωτήπων να δεχθούν ότι, μπορούν να ότι μπορούμε να κάνουμε συστάσεις και να δέχονται να αλλάζουν εξ άντε εκ των προτέρων τις μακροοικονομικές πολιτικές τους ώστε να υπάρχει μια διεθνής οικονομία όσο ανθεκτικότερη γίνεται και που μπορεί να μας δώσει αυτό που όλοι θέλουμε ανάπτυξη, βιώσιμη ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, βιώσιμες θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο κοινός μας στόχος τελειώνουμε με αυτόν τον τελευταίο νομισματικό διάλογο αυτή εδώ τη πενταετία του Κοινοβουλίου. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να σα ευχαριστήσω γιατί οφείλετε να έρθετε. Είναι φυσιολογικό λοιπόν να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ταυτόχρονα όμω θεωρώ ότι είχαμε μια πολύ καλή αμοιβαία σχέση, χρήσιμη, η οποία πρέπει να προχωρήσει κι άλλο. Ξέρω ότι οι συνάδελφοι αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στο πώ ασκούμε αυτή την ευθύνη, την ευθύνη μας και το μάτι αυτό τι συμβαίνει στην Ευρώπη και στην Αμερική όπου η κατάσταση δεν είναι πάντα συγκρίσιμη αλλά στο νομισματικό αυτό διάλογο πρέπει να κρατάμε σταθερά τη θέση στο μεταρρύζι μας. Χαίρομαι λοιπόν γι' αυτό. Σας, ευχαριστώ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλοι θα περιμένουμε με ανυπομονησία τα πορίσματα των J20 που απέδειξε ότι το θέμα που θα χειριστεί είναι μια σοβαρή πρόκληση για τη διεθνή οικονομία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ